So, hello, good morning. Καλημέρα σας. Ε, δεν είμαστε και πολύ παρόντε. Oh, this is a great day. Αλλά θα αρχίσουμε. Ε, είναι για μένα πολύ σημαντική ημέρα, γιατί καταρχήν προεδρεύω εδώ, ως αντιπρόεδρος του αντιπρόεδρου, τόσο πάντων. Αλλά κύριε Σερδαπικοστή, ε, επέτειος γενεθλίου του Bob Dylan. Some kind of I wish I could say that Thames... Ε, άλλαξαν οι καιροί, αλλά άλλαξαν και οι καιροί και για την ενιαία αγορά. Από τη μία έχουμε τους ε, Rolling Stones, από την άλλη μεριά έχουμε I'll go my way για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Μπομπ να μπορεί να κάνει ένα σφάλμα και εμείς στην συζήτηση για την ενέργεια επίσης μπορούμε να κάνουμε ένα σφάλμα. Uh, adoption of draft agenda. It has been distributed. Uh, Έχετε πάρει την ημερησία διάταξη. Αν δεν υπάρχουν διαφωνίες, παρατηρήσεις, μπορούμε να την εγκρίνουμε. This meeting is being web streamed. Welcome to all who are watching us online. τα μέλη της ΣΥΜΚΟ έχουν κληθεί να πάνε στις 3 ώρα το απόγευμα στη συνεδρία της Επιτροπής ΕΝΒ για μια παρουσίαση για τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. Δεν θέλω να καθορίσω καλωσορίζω την κυρία Πρέντεργκάς που είναι καινούρια εδώ και ανικασιστά, τον άλλον Κέλλη που είναι τώρα ε, υπουργό. Σας καλωσορίζουμε θερμότατα λοιπόν. Τι άλλο έχουμε εδώ. Έγκριση των πρακτικών. Σημείο 3. Το συνεδριάσιο στις 16 Μαρτίου, 1 η και 22 Μαρτίου Μαρτίου και 11ης έως 13 η Απριλίου. Αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις θα τις κάνετε παρακαλώ μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα πάμε στα κυρίω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα είναι η επίσκεψη στην Πολωνία και είχαμε εδώ κάποιον που ήταν παρόν και θέλει να μας παρουσιάσει τα σχόλιά του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να περιμένω λιγάκι, νομίζω. Για να βάλουν όλα τα ακουστικά τους και να γυρίσουν στη σωστή γλώσσα. Κάναμε μια πολύ χρήσιμη επίσκεψη στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα. Στην Κρακοβία ξεκινήσαμε. Εγώ, μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ολλανδία, πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο να δει κανένα τέτοιο ενθουσιασμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κρακοβία μιλήσαμε με επιχειρηματίες που όλοι εξυμνούσαν την εσωτερική αγορά μία ανησυχία, όμως για διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Οι εξαγωγές από την Πολωνία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποφέρουν λόγω των διαφορετικών φόρων, ιδίως όσον αφορά το ύψος του ΦΠΑ. Το ύψος του φόρου βέβαια είναι θέμα των κρατών μελών και το πιο αναχρονικό είναι η δομή των φόρων. Από την που πήγαμε στη Βαρσοβία που συζητήσαμε με την Μενοντική Πολωνική Προεδρία συζητήσαμε με έναν ενθουσιώδη υφυπουργό θεμάτων Ευρώπης και εσωτερικής αγοράς. Συζητήσαμε επίσης και στο Κοινοβούλιο και στη Βουλή και στη Γερουσία είχαμε συνομιλητές και εξετάσαμε διάφορα θέματα ΙΜΚΟ. Και εκεί υπάρχει επιθυμία όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική υπογραφή και το θέμα της κυρίας Ρούλε όσον αφορά τις ε, δημόσιες αγορές να προχωρήσουμε κάποιο πιο γλίγορα. Η πολωνική οικονομία αυξάνεται γλίγορα και συνεχώς. Και θα θέλα να εκμεταλλευτούν την Προεδρία τους ε, του Συμβουλίου για να προχωρήσουν και να προωθήσουν θέματα της ΣΥΜΚΟ. Ευχαριστώ τους οργανωτές, ευχαριστώ όλους από τη γραμματεία της ΣΥΜΚΟ γιατί όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα και πολύ καλά. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Φανεκάμ. Κατά βάση η ημερησία διάταξη αρχίζει με τη δική σας έκθεση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Μποπτήλαν ε, ήταν και επίση μοτοσυκλετιστής. Νομίζω ναι, κάπου τον είδα σε μια φωτογραφία με μοτοσυκλέτα που φαίνεται. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο γιατί έχω κάποια σχόλια για το θέμα αυτό της έκθεσής μου. Ε, έχετε πάρει την έκθεση αυτή στα χέρια σας, νομίζω. Ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν σε αυτή. Είναι πολύ βαριά εργασία να προετοιμάσει κανένα μια τέτοια έκθεση. Δεν το είχα φανταστεί ότι θα ήταν τόσο δύσκολο. Αλλά ε, και στην ε, γραπτή μετάφραση του κειμένου και στην εκτύπωση υπάρχουν κάποια σφάλματα γιατί οι τεχνικές προδιαγραφές των Enduro και του Flyer έχουν αντιστραφεί. Μπορούμε να το διορθώσουμε όμως με μια τροπολογία. Και όσον αφορά τις μικρές σειρές, παράρτημα 3, και εκεί υπάρχουν προβλήματα αριθμών. Κατηγορία L1, Α1, Β και Γ θα έπρεπε να λέει αναγράφεται 50, όχι 20 και στην επόμενη κατηγορία 100 αντί 50. Κάναμε όλες τις τροπολογίες για τα παραρτήματα ήδη και οι συνεργάτες μου προέτοιμασαν. το πήρατε κυρία Βέλου. Το καινούριο το κείμενο το έχετε. Ωραία. Το καινούριο παράρτημα λοιπόν έχει διανεμηθεί ήδη και συμπεριλαμβάνει όλες τις τροπολογίες και έτσι είναι πιο ευανάγνωστο το κείμενο προφανώ. Όσον αφορά το περιεχόμενο τώρα, κύρια Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Έγιναν οι απαραίτητε συζητήσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή της πρόταση τη Κομισιόν. Για διάφορα σημεία διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή και για μια σειρά κατηγοριών ε, έχουμε συμπεριλάβει περισσότερα ε, περισσότερα οχήματα, δηλαδή Enduro S1, Trial S2 και ATV, ε, ATV έχουν συμπληρωθεί τις κατηγορίες αυτές και αυτό γίνεται νομίζω γενικά καλά δεκτό. Μετά προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε, να απλουστεύσουμε αν θέλετε το χρονικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύπλοκο. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μόνο τρία στάδια, όχι οκτώ όπως είπαν, υπήρχαν αρχικά. Οι αντιδράσεις μέχρι στιγμή ήταν θετικέ. Από την Κομισιόν ανεπίσημα ακούσαμε ότι όσον αφορά τις εκπομπέ θα πρέπει να παραμείνει ένα ενδιάμεσο στάδιο. Και θα αναφερθώ σε αυτό, στο θέμα του περιβάλλοντος δηλαδή. Είναι και αυτό σημαντικό en Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα δίτροχα ε, μολύνουν την ατμόσφαιρα αρκετά. Δεν χρησιμοποιούν τόσο πολλά, αλλά οι εκπομπές ανά χιλιόμετρο είναι ε, πολύ σημαντικές. Το παραδέχομαι, τι να κάνω. Βέβαια εδώ είμαι τώρα ως ε, εισηγητής και όχι μοτοσυκλετιστής. οι Γερμανοί και άλλοι χριστιανοδημοκράτες παρακολουθούν στενά την, ε, την έκθεση αυτή θα έλεγα. Μετά τα συστήματα διάγνωσης και δεν ξέρω κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο και για τα μικρά ε, οχήματα και τα μοτοποδήλατα. Αλλά θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα υπάρχουν και τροπολογίες. Είμαι σίγουρος. Περνάω τώρα στα μέτρα ασφαλείας, Πρόεδρε. Ε, είχαμε μια καλή συζήτηση στο Κοινοβούλιο και με το συναδέλφους της Επιτροπής Τραν για το θέμα κατά πόσον όλα τα συστήματα τροχοπέδησης, ΕΜΠΕΣ και ABS, θα πρέπει να επιβληθούν για όλα τα μικρά δίτροχα. Εγώ καταρχήν είμαι κατά, αλλά αισθάνομαι την πίεση να το συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Το θέμα είναι όμως ποιο θα είναι το όφελο αυτό για απλά μοτοποδήλατα και για σκούτερ. Δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο και γι' αυτό δεν ξέρω κατά πώς θα πρέπει να επιβάλλουμε αμπές. και αυτό είναι ένα προσυζήτηση θέμα. Οι τροπολογίες ε, των ε, μοτοσυκλετών, ε, οι τροποποιήσεις μάλλον στις μοτοσυκλέτες είναι δυνατές. Υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται μόνο κάνουν κάποιες αλλαγές, πιο ισχυρές μηχανές κλπ. Αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε, αλλά στους λεγόμενους free riders θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να κάνουν κάποιες αλλαγές στις μοτοσυκλέτες τους. Τώρα θα πρέπει να εξτάσουμε το θέμα των μικρών επιχειρήσεων που θέλουν να κατασκευάζουν μικρές σειρές μοτοσυκλετών ή διτρόχων. Και θέλαμε η Κομισιόν να προσαρμόσει την πρότασή της για να μπορούν και αυτές οι μικρές σειρές να εγκρίνονται όσον αφορά τους τύπους. Και υπάρχει κάτι άλλο μικρό. Το θέμα της πρόσβασης στις πληροφορίες για ε, συντήρηση και επισκευές. Δεν θέλουμε δηλαδή οι κατασκευαστές να μην δίνουν τις πληροφορίες αυτές ούτε στους εμπόρους ούτε στους καταναλωτές. Προσπαθήσαμε λοιπόν η πρόσβαση αυτή της πληροφορίας να είναι κατά δυνατόν ευρεία. Όσον αφορά την προετοιμασία της έκθεσης αυτής, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι οργανώσαμε και μία ακρόαση σχετικά, η οποία έτυχε έντονης ε, συμμετοχής μέσω και του web streaming και κάναμε και κάποιε επισκέψεις. Πήγαμε στην Πολόνια, στο Ντουκάτι, στην τη Βέκιο, και είδαμε εκεί την ε, ε, εταιρεία κατασκευής ε, των σκούτερ και πήγαμε και στο Έσεν, στο ΤΥΦ Και τώρα θα επισκεφτούμε και μία μονάδα παραγωγής Honda και BMW. Αρχές Ιουλίου νομίζω θα γίνει αυτή η επίσκεψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές, οι οποίοι ανεπίσημα πολλά σκεφτήκανε και επίσημα φαντάζομαι θα μου το πούνε τώρα για να ξέρω τι σκέφτονται. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Φαντενκάμπ. Είμαι σίγουρη ότι μέσω του web streaming πολλοί μοτοσυκλετιστές ε, παρακολουθούν την συνεδρίαση αυτή και χαίρομαι που κάνατε αυτές τις παρατηρήσεις. Έχω πρώτα ε, γεγραμμένου στο κατάλογο των αγοριτών τους ε, σκιώδεις εισηγητές, Κριστίν Βέστφαλ. Ja, guten Morgen, sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr verehrter Herr Berichterstand. Καλημέρα σας. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά φωνεκά εγώ δεν είμαι αυτοσυγκρίστρια, αλλά παρόλα αυτά ε, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και νομίζω και εγώ και οι συνεργάτες μου τις τελευταίες εβδομάδες πολλά έμαθαν και για τους μοτοσυκλίτσες, αλλά και για τα δίτροχα και τρίτροχα οχήματα. Καταρχήν εισαγωγικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς ε, κύριε Φανενκάπ τόσο δεσμευμένος ήσασταν για τη συζήτηση για το θέμα αυτό και για την έκθεσή σας. Σε πολλά σημεία μπορούμε να την υποστηρίξουμε, αλλά όπως είπατε και εσείς, όχι σε όλους εμείς. Θεωρώ πολύ θετικό ότι διαβρύνατε το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία στα ATV και Enduro. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ καλό για την εργασία μας στο μέλλον. Ε, έχω όμως διαφορετική άποψη όσον αφορά τη σημερινή εισαγωγή των ευρωπροδιαγραφών. Mm. Νομίζω ότι η παράγραφο 3 αντικατοπτρίζει την ε, πραγματικότητα. Γιατί όλα τα οχήματα σχεδόν βρίσκονται αυτή τη στιγμή τεχνολογικά σε αυτά τα πρότυπα. Όπως είπατε και εσείς, ε, νομίζω ότι αυτό που προτείνεται αυτή τη στιγμή και από την Κομισιόν αλλά και από εσά δεν είναι και πολύ φιλόδοξο. Δηλαδή, εάν η Euronorm 4 και 5 συνενωθούν στην ημερομηνία εισαγωγή ε, της Euronorm 4, δηλαδή το 2015. Αυτό θα μου φαίνεται ε, πάρα πολύ θετικό. Το ίδιο ισχύει και για το ότι ίσως μια σταδιακή εισαγωγή θα ήταν καλή, αλλά γιατί να εξαιρούν από το ΕΠΕΝΤΕ τα μοτοποδήλατα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θέλουμε να απαγορεύσουμε τη δυνατότητα τροποποίησης των ε, οχημάτων αυτών και το ΟΠΕΝΤΕΙ μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ελέγχου. Mm. Και γιατί, γιατί να επιτρέψουμε να γίνονται κάποιες αλλαγές από τους χρήστες και δεν σας μιλάω εδώ στην μητέρα ε, δύο κορών, 9 και 13 ετών που δεν θέλουν να τα Αυτό για μένα είναι θέμα ασφαλείας. Το συνδυασμένο σύστημα τροχοπέδησης δεν είναι εναλλακτική στο σύστημα ABS, anti-block. Ίσως θα πείτε ότι θα υπάρξει τελικά ε, μια εκαθάριση αν θέλετε στην αγορά εάν το ABS γίνει υποχρεωτικό για τα δίτροχα και τίτροχα και δεν θα υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα. Αυτό για μένα δεν είναι ε, επιχείρημα. Ναι, κάποια οχήματα θα εξαφανιστούν, κάποιοι τύποι οχημάτων, αλλά όχι οι κατασκευαστές ήδη, γιατί εδώ συζητάμε για τη δυνατότητα μέσω ενός κανονισμού να μειώσουμε τον αριθμό των νεκρών από δυστυχήματα με τα οχήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι μπορούμε να δεχθούμε αλλαγές στο design και την εξαφάνιση κάποιων τύπων ίσως των οχημάτων. Είμαι πεπισμένη όμως για την δημιουργικότητα και τη δυνατότητα καινοτομίας της σχετικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Γιατί τελικά μπορούμε και στα παιδικά κάρτ να εισαγάγουμε τα συστήματα αυτά τροποπέδησης anti-block ABS. Η τιμή δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί μάλιστα να υπάρχει και μείωση της τιμής εάν υπάρχουν λιγότεροι τύποι οχημάτων που κατασκευάζονται. Είμαι σίγουρη ότι θα πετύχουμε τις επόμενες εβδομάδες να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και τελειώνοντας, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Φανακάμ, κύριε Σιγητά, για την καλή σας συνεργασία και τις επισκέψεις εργασίας επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βέστφαλ. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, Μάντες δεν εδώ, Κρότσμαν εσείς. Ναι, ο κύριο Μάντερ είναι υπεύθυνο ε, στην ομάδα μα, που δεν είναι εδώ και δεν θέλω να το σχολιάσω. Ωραία. Ο κύριο Άμπερ δεν είναι εδώ, η Χάρη Ρίλε. Τα ακουστικά μου δεν λειτουργούν, αλλά το μικρόφωνο φαίνεται ότι λειτουργεί, οπότε κάτι είναι αυτό. Θα ήθελα σε ορισμένα σημεία να συμφωνήσω με την προλαλή σα. Ή μάλλον να αρχίσω με το σωστό, με τι ευχαριστίε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο εισηγητή πραγματικά συνεργάστηκε παραδειγματικά με εμά του σκιώδες εισηγητέ και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Ο τρόπος εργασίας ήταν απόλυτα διαφανή και μα βοήθησε βήμα προ βήμα να προχωρήσουμε. Δεν μπόρεσα να πάω σε όλε τι επισκέψει. Παρ' όλα αυτά ήμασταν πάρα πολύ ενήμεροι και θα ήθελα να πω ότι αυτό που προετοιμάστε τώρα είναι ευνόητο και σε γενικέ γραμμέ μπορώ να το υποστηρίξω. Πραγματικά κύριε Φανεκόπ η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Σε ένα σημείο με το οποίο θα ήθελα να συμφωνήσω με την προλή σα είναι το θέμα των εκπομπών όπου κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο φιλόδοξοι. Αυτό δηλαδή για την Euronorm 4 και 5 νομίζω ότι θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Τώρα κατά πόσον θα τη συνενώσουμε. Είναι καλό, αλλά θα πρέπει και η χρονική στιγμή που θα επιλεγεί να είναι επίσης θετική. Ένα αυτό. Δεύτερον, προσωπικά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την τροχοπέδηση αντιμπλοκ ABS να είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα μοτοποδήλατα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, γιατί έχω κάποιες αφιβολίες. Το πρόβλημά μου είναι αλλού και θα πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εξελίξεις στον τομέα των διτρόχων, τριτρόχων και τέτρατρόχων αυτή τη στιγμή επιταχύνεται και υπάρχουν όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά οχήματα στην αγορά και η εξέλιξη δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Παραδείγματος χάρη έχουμε τα 5LX, δηλαδή τα ηλεκτρονικά ποδήλατα με υποστήριξη κινητήρα. Τι θα μας ενδιαφέρει, το θέμα της ισχύω εκεί θα βασιστούμε στον ορισμό ή όσον αφορά την ταχύτητα. Γιατί εάν τα εγκρίνουμε αυτά ε, μέσα στην πόλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε διαφορετικού τύπου οδηγούς. και θα πρέπει η ταχύτητα να είναι διαφορετική από την πόλη, στην Ήπεθρο κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει νομίζω να συζητήσουμε. Και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε κάποια ρήτρα αναθεώρησης. Γιατί βλέπουμε ότι οι τάσεις είναι προς τον ηλεκτρικό τομέα των οχημάτων. Και αν εμείς ε, ορίσουμε όρια μέσα στον ορισμό των τύπων, ίσως παρεμποδίσουμε την εξέλιξη. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Ίσως θα ήταν καλό μαζί σας και μαζί και με την Κομισιόν να εξετάσουμε τι θα γίνει. Γιατί όταν προετοίμαστε την πρόταση της Κομισιόν, αυτή η εξέλιξη που βλέπουμε σήμερα δεν προβλέπεται. Και σε δύο χρόνια θα έχουν επίσης αλλάξει τα πράγματα. Θα ήταν λοιπόν καλό να έχουμε μια ρίτερη αναθεώρηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάντες είναι εδώ και επομένως Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Ναι, έχω κάποια σχόλια να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έφτασα αργά, αλλά χωρίς καφέ δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έπρεπε να τον καφέ μου. Συγγνώμη, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον ε, Βιμ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ανοιχτός ε, ε, στη συνεργασία μαζί μας. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ήδη έχουν υποθεί. Σχετικά με το 13, περιορισμένος αριθμός ε, ε, οχημάτων, εκεί χρειάζεται κάποια περαιτέρω αποσαφήνιση. Δηλαδή τι σημαίνει περιορισμένος αριθμός, τι εννοούμε με περιορισμένο αριθμό κλπ. Τι άλλο, τι άλλο. Συμφωνώ με τις υποκατηγορίες αλλά βεβαίω θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο πιο στενά το τι σημαίνει η εισαγωγή ειδική κατηγορίας και εδώ χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση, όμω η γενικότερη προσέγγιση είναι πολύ καλή. Μιλήσαμε για συμμόρφωση των ε, οχημάτων και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε και την αμοιβαία αναγνώριση συστημάτων ε, τα κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε όλες τις χώρες. Άψογα, το περάσαμε και αυτό λέει ο μιλητής. Προχωρούμε. 15 ε, αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να μιλήσουμε για ε, ε, ε, δραστηριότητες ψυχαγωγικές καθαρά από τη μία πλευρά και το διαγωνιστικό κομμάτι από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί δηλαδή αυτό. Εάν είναι δυνατόν, θα ήθελα να προσθέσω και το έχω ήδη συζητήσει με το Βίμ. Πιστεύω ότι η ορατότητα ε, η πλευρική είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι εδώ, δηλαδή να έχουμε κάποιους καθρέφτες, πλαϊνούς κτλ. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε μοτοποδήλατα τα οποία εμπλέκονται σε ατυχήματα γιατί πολύ απλά το αυτοκίνητο, το μεγαλύτερο όχημα δεν είδε το μοτοποδήλατο ή το μηχανάκι. Επομένως ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βελτιωθεί η ορατότητα αυτών των δικύκλων ε, εναρμονισμένες απαιτήσει ε, αδειοδότησης. Ναι, υπάρχει μια ειδική οδηγία επ' αυτού, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι και για τα μοτοποδήλατα θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ενιαία αδειοδότηση. Ναι, βεβαίω, όταν μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα φυσικά θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, φόρτιση σε διάφορα σημεία ε, και θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα ανταλλαγής ε, μικρών, μικρού όγκου ορευτών μπαταριών έτσι ώστε να μην χρειάζεται κανεί να κουβαλάει την μπαταρία του μαζί και όταν πέσει η ισχύ της του να μπορεί τουλάχιστον ένα κομμάτι, να το φορτίσει, να το ανταλλάξει. Ναι, λέω απλώς ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Γιατί είναι γεγονός ότι εμείς δημιουργούμε προϋποθέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά η βιομηχανία είναι αυτή η οποία μέσω των καταλήλων μέσων και ε, ρυθμίσεων θα πρέπει να δώσει λύσεις. Um, uh, Τελευταίο, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ασφάλεια των εποχουμένων κάθε πέντε χρόνια να γίνεται ένας τεχνικός έλεγχος, ο οποίος θα γίνεται όμως από επίσημο φορέα ε, και θα διέπεται από την, θα οργανώνεται, εν πάση περιπτώσει, από το κράτος, ε, θα, να υπάρχει μια, ένας κατάλογος για αυτό το check-up, για αυτόν τον έλεγχο, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι κάθε πέντε χρόνια ελέγχονται τα πάντα. Πιστεύω ότι είναι ε, σωστό να γίνεται αυτό έτσι ώστε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος να ξέρει ότι ε, είναι εντάξει και ότι μπορεί να λειτουργήσει καλά το όχημά του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σουάπ, παρακαλώ. Θέλετε κάτι να πείτε, κυρία Ρούλε? Do you want to say Τώρα. Point amendment 65. Για την τροπολογία 65 έχω μια ερώτηση. Ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως. Α, να μιλήσω γερμανικά καλύτερα. Αναφερθήκατε στα, στα μέτρα ε, που αναφέρουν διαφορετικά για τον, τους διάφορους τύπους δεν ξέρω γιατί το κάνε, κάνετε αυτή τη διάκριση για μεταφορά επιβατών, μεταφορά επιβα, ε, εμπορευμάτων διαφορετικά. Ευχαριστώ, με συγχωρείτε κύριε Σουάμ. Νομίζω ότι, νόμιζα εγώ ότι ήταν σχόλιο για τα αυτά που είπε ο κύριος Μάντες. Ευχαριστώ. Και εγώ έβαλα στο γάλα στο καφέ μου να το πιω. Εντάξει, όλοι έτοιμοι. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Φαντεγκάρ γιατί εργάστηκε πάρα πολύ προσεκτικά σε αυτή την τόσο τεχνική οδηγία και τα κυριότερα σημεία που αναφέρθηκαν ε, διευκρινίσαν νομίζω ικανοποιητικά και υπάρχουν και πολλές δυνατότητες συμβασμών. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ, αλλά δεν μπορώ να το εκτιμήσω ιδιαίτερα και δεν με βοήθησε και η συζήτηση που έγινε μέχρι στιγμής είναι το θέμα του εξοπλισμού με συστήματα τροχοπέδησης ABS, anti-blocking. Γιατί νομίζω ότι η ασφάλεια των οχημάτων αυτών, ιδίω για τους νέους, δεν είναι τόσο καλή, δεν έχουν δηλαδή συμπεριληφθεί όλες τις δυνατότητες ε, οι τεχνικές στα οχήματα. Απ' την άλλη μεριά βέβαια αν συμπεριλάβουμε τα πάντα Πολλοί από τους νέους δεν θα έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να αγοράσουν τα οχήματα αυτά. Και θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε εσείς κύριε Σιγητά την διάκριση και την αξιολόγηση των στοιχείων οικονομικών αφενός και ασφάλειας αφετέρου. Ευχαριστώ. Okay, Mr. Θέλετε να απαντήσετε τώρα, κύριε Φαντερκάμπ, ή να περιμένουμε και την Επιτροπή. Θέλετε... Νομίζω μετά, αφού πάρει το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μαρτίνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Madam Chair, and... Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Uh, Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Βάντερ για την εξαίρετη εργασία που έκανε και η οποία έγινε και με στενή συνεργασία και με μας, με πλήρη διαφάνεια, όπως άλλωστε σημείωσαν και πολλοί ε, των προλαλισάντων και βεβαίως ε, ε, είχε, έδωσε την δυνατότητα καλή συνεργασίας πάνω και σε πολιτικά αλλά και σε τεχνικά ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ για τη στάση του τον εισηγητή όσον αφορά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα τρία στοιχεία τα οποία ε, αναφέρθηκαν από τον κύριο Βάντεν Κάπ και, και από τους βουλευτές όσον αφορά την κατηγοριοποίηση. Ε, βεβαίως ε, είμαστε ανοιχτοί και καλωσορίζουμε το γεγονός ε, ότι ε, έχουμε πιο λεπτομερείς κατηγορίες γιατί αυτό μεταξύ άλλων θα μας δώσει την δυνατότητα καλύτερης στοχοθέτησης των κατηγοριών των οχημάτων όσον αφορά την ασφάλεια και κυρίως όσον αφορά το ζήτημα της εισαγωγής ε, του ε, ABS και γενικότερα προηγμένων συστημάτων πέδησης ε, είναι γεγονός ότι εδώ έγινε μια προσπάθεια να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και του κόστους. όσον αφορά την καθυστέρηση εισαγωγή προηγμένων συστημάτων πέδησης κατά ένα χρόνο, αυτό δεν οφείλεται μονάχα στο ε, κόστος, ε, αλλά και στο ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο ε, μέχρι ότου όλοι να αποκτήσουν το σύστημα αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυξάνονται τα ατυχήματα και μάλιστα τα θανατηφόρα όσον αφορά του μοτοσυκλετιστέ. Εμείς προ προτείναμε κάτι τέτοιο γιατί ξέρουμε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο όσον αφορά ε, την θέση σε ισχύ νέων ε, ε, στοιχείων και το να θεσμοθετήσουμε την 1η Ιανουαρίου του 2017 για την ε, υποχρεωτική εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων πέδησης σε κάθε είδος ε, διτρόχου ε, πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην ασφάλεια αλλά προϋποθέτει ότι θα έχουν λυθεί κάποια προβλήματα. Στο επόμενο σημείο θα ήθελα να πω ότι ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το πρώτο σημείο γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή πριν από το 2017 δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα και όλα τα στοιχεία όμως έχουν πλέον ε, συλλεχθεί ε, και καταδεικνύουν ότι όχι μονάχα είναι σημαντικό να καθορίσουμε φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τις εκπομπές αλλά ότι και ο χρόνος που θα γίνει αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε, κατά 62% συμβάλλει η κατηγορία αυτή ε, στις ε, εκπομπές τέτοιου είδους αέριων και επομένως καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να να βελτιωθεί η κατάσταση. Πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο να έχουμε τέτοια στοιχεία κυρίως ε, όσον αφορά τις εκπομπές σε μικρές αστικές ε, περιοχές. Πιστεύουμε ότι εάν διατηρήσουμε ε, την προσέγγιση του πρώτου στόχου, τότε θα είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Όσον αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα να πω ότι και κάποιες χώρες μέλη Επίσης έχουν σε μερικές περιπτώσεις εισάγει ε, κάποια μέτρα απαγόρευσης των ε, ακόμα και των μικρών ε, σκούτερ από τον εσωτερικό δακτύλιο των μεγάλων πόλεων και Ε, πιστεύουμε ότι μια γενικευμένη χρήση των διτρόχων θα μπορούσε ε, να διευκολύνει σε πολλές περιπτώσεις ε, την κυκλοφορία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καλωσορίζουμε κάθε προσπάθεια για, νέ, για εισαγωγή νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να δοθούν νέες λύσεις και ώστε μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας να ανοιχτούν κάποιες δίωδοι για νέες τεχνολογίες τεχνολογίες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα οχήματα ε, θα είναι πολύ ασφαλή και όσο γίνεται περισσότερο ε, φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και ότι θα είναι τουλάχιστον όσο ασφαλή όσο είναι όλα τα άλλα οχήματα. Ε, όταν αρχίσουμε βέβαια να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά ε, τις κατηγορίες βάση του βάρους, ε, όντως φτάνουμε και στο πρόβλημα των μπαταριών και αυτό είναι ένα μειονέκτημα όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα δίκυκλα. Πάντως η θέση μας είναι ότι πρέπει να προωθήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βαντενκάπ να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε πολύ, αλλά ε, τα πράγματα θα γίνουν λίγο πιο τεχνικά τα επόμενα 10 λεπτά. Πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ε, αυτό είναι απαραίτητο γιατί η έκθεση είναι επίγουσα. Θέλω να συγχαρώ την πολύ καλή συνεργασία, την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τους σκιώδεις συζητητές και να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Υπάρχουν μεν διαφωνίες, αλλά η διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ε, θα ακολουθήσω την ίδια ε, προσέγγιση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, καταρχάς, στην εισαγωγή που σας έκανα, παρότι πραγματικά είμαι φανατικός των ε, δίτροχων, έχω πιστεί ότι μπορούν να ρυπάνουν παρόλα αυτά την ατμόσφαιρα. Και πραγματικά είμαι διατεθειμένος να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτό. Το έχουμε πει με τους σκιώδεις, θα ξαναμιλήσουμε για τις ημερομηνίε, αλλά θα ήθελα και για τον κλάδο. Θα ήθελα να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο τομέα των αντιτρόχων. Υπάρχει μια βαθιά οικονομική κρίση, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο κλάδος, η βιομηχανία νομίζω ότι ε, ακροάζεται και ίσως ε, καταλαβαίνει τι γίνεται και μπορεί κάτι να γίνει. Τώρα με τους άλλους κλάδους θα έπρεπε επίσης να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. De tweede opmerking van mevrouw Westphal over de... Παρατήρηση της κυρίας Βέστφαλ για τα σκούτερ και για τα διαγνωστικά συστήματος, ε, συστήματα οχημάτων. Αυτά πράγματι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο. Υπάρχουν πιο αυστηρές διατάξεις και σε ό,τι αφορά τον κινητήρα και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως και τον παράγοντα κόστος. Ένα σκούτερ 1.200 ευρώ ε, δεν μπορεί να έχει και έναν εξοπλισμό αξίας 400 ευρώ, δεν είναι εύκολο. Και σε ό,τι αφορά το σύστημα πέδησης, ένας νεαρός ή μια νεαρή 16 ετών μπορεί να οδηγεί σκούτερ που έχει αυτό το σύστημα ή ένα αυτοκίνητο που έχει αυτό το σύστημα, αλλά δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ξέρει και να το χρησιμοποιήσει. Και οι νέοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων. θα δούμε και με την Επιτροπή Μεταφόρων πώς μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την πρότασή μας για τον τομέα αυτό. Αλλά θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι γίνονται όλο και πιο φθηνά αυτά τα συστήματα, χρόνο με το χρόνο. Η Harley Davidson ακόμα ζητά 1.200 ευρώ για τα συστήματα αντιεμπλοκής. 600 ευρώ κέρδος για την ε, Harley. Ε, εντάξει, θα δούμε και πώς εξελίσσεται. Αυτό μας λένε ότι μπορεί να κοστίζει 800, 80 ε, ευρώ μάλλον, ε, αλλά για να τοποθετηθεί ε, πάνω σε ένα ε, μηχανάκι μπορεί να έχει κόστος εργατικά 200-300 ευρώ. Θα τα δούμε αυτά. Καταλαβαίνω όμως αυτά που λέει η κυρία Βέστφαλ για τις εκπομπές, για τα διαγνωστικά συστήματα οχημάτων και για τα συστήματα πέδησης. Ε, κυρία Ρούλια τώρα. συμφώνησε με τις παρατηρήσεις αυτές. Κυρία Πρόεδρε, τα ηλεκτρικά ποδήλατα ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχω συζητήσει με υποστηρικτές αυτών των ε, οχημάτων, αυτών των δικύκλων, αλλά και με τους κατασκευαστές τους, οι οποίοι θα ήθελα να υπάρχει λόγος μεν για περιορισμό των επιδόσεων, αλλά Παρ' όλα αυτά, αυτά τα ποδήλατα μπορούν να φτάσουν σε μεγάλες ταχύτητες και νέοι και πιο μεγάλοι. Ε, μπορούμε να τους δούμε να κατεβαίνουν ένα ε, λόφο 45 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς να φοράνε καν κράνος και να μην έχουν καμία άλλη προστασία. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε, να μιλήσουμε και με τον κλάδο για αυτό το θέμα. Το θέμα επίσης ε, των ε, δικύκλων, τρικύκλων και τετρακύκλων με ηλεκτρική προώθηση. Συμφωνώ με την κυρία Ρούλη ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε τις τεχνικές εξέλιξη, τεχνική πρόοδο. Πάντοτε όμως πολύ γρήγορα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ζήτημα του βάρους. Τα οχήματα αυτά είναι αρκετά βαριά λόγω των, ε, συστημάτων συσσωρευτών των μπαταριών που υπάρχουν σήμερα αν κάποιος ε, εφεύρει μία μικρή μπαταρία, αυτό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Οπότε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα μπορούσαν πλέον να αναπτυχθούν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Ε. Αλλά έχουμε το θέμα του βάρους για αυτά τα οχήματα. Και δεν νομίζω ότι η οδηγία για τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα συστήματα. Συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία Ρούλε. Οι τεχνικές εξελίξεις, η τεχνική πρόοδος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να ληφθεί και στη συγκεκριμένη διάταξη. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 65, πάντα ε, στην κυρία Ρούλη αναφέρομαι, Έχουμε και μία συνέντευξη που λέγεται ρόλια και γι' αυτό το ρίλε ρόλ περδεύομαι. Χάιντι, ε, με 65. Θα σας λέω κυρία Χάιντι για να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία Χάιντι, για να είναι πιο απλό. Χωρίς κυρία Χάιντι, εντάξει. Λοιπόν, Χάιντι. Μιλάμε για τη μεταφορά εμπορευμάτων. με όχι πολύ μεγάλο βάρος, αλλά έχουμε και κάποια άλλα οχήματα που μεταφέρουν λίγο πιο βαριά εμπορεύματα και έχουν και ένα αποθηκευτικό χώρο. Αν ανεβούμε ε, στην κατηγορία των κιλών μέχρι 700 κιλά, τότε πρέπει να αλλάξουμε κατηγορία. Έχουμε την κατηγορία M. Τώρα, τροπολογία 50, Μάντελς. Λέγαμε στον κύριο Μάντελς. Αθλητικές δραστηριότητες. και στο δρόμο αλλά και παντός εδάφους off-road. Δεν θα, να υπάρχουν, δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί για τα οχήματα που, δημιουργούνται, που χρησιμοποιούνται σε αθλητικές δραστηριότητες, αγώνες, ταχύτητας κτλ. Δεν έχουμε πολλά πρόβληματα με τα συστήματα πέρυσι εκεί. Ε, Τέλο πάντων θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την πλευρική ορατότητα των μηχανών, θα τα κάνουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα τις μηχανές. Δεν μπορούμε να τα παραφορτώσουμε. Ε, βέβαια, σίγουρα η ασφάλεια ε, στην κυκλοφορία των μηχανόβιων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, οι ηλεκτρικές, ε, μάλλον τα ηλεκτρικά οχήματα και οι μπαταρίες που μπορούν να επαναφορτίζονται και η ομοιομορφία που θα πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα σημεία. Έχουμε διάφορες, ε, διάφορα δελτία τεχνικά, άλλο για χαμάχα και άλλο άλλες εταιρείες και αν δεν υπάρχει ομοιογένεια και ομοιομορφία τότε θα έχουμε προβλήματα. Επίσης ε, υπάρχει μια πρόταση για την ε, έγκριση ε, που θα πρέπει να δίνεται κάθε πέντε χρόνια. Βέβαια, παρότι κατανοώ, δεν είμαι υπέρ. Δεν νομίζω ότι περισσότεροι μοτοσυκλετιστές κάνουν αιτήσιο σέρβις. Είναι ένα θέμα πολύ λεπτό Πρέπει να υπάρχει ένα είδος υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου. Μετά τις παρατηρήσεις που έκανα απευθύνω στις κυρίες Βέσταλ και Ρούλη, νομίζω ότι έχω απαντήσει και στα σχόλια του κυρίου Σβάπ. Χθες εξεφράστησαν τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και θα δούμε και τι θα πούν και για τα συστήματα πέδησης και για τα διαγνωστικά συστήματα. Θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για, την, ε, για τις τροπολογίες είναι 20 Ιουνίου. Και θαύμα. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Yeah, good. Wonderful. Um... Uh, Ακεραιότητα και διαφάνεια της αγοράς ενέργειας. Έχετε τις ε, κάρτες ε, ψηφοφορίας. Ραφάλ Τσαρκόφσκι. Πολύ σύντομα κυρίες και κύριοι. Έχουμε προετοιμάσει γνωμοδότηση για την ακαιρεότητα και διαφάνεια της αγοράς ενέργειας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγητές για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε επ' αυτής της γνωμοδότησης. Ε, αρχικά έπρεπε να αποφασίσουμε τι θέλαμε να συμπεριληφθεί στην γνωμοδότηση αποφασίσαμε να συστάλλουμε λίγο το πεδίο έτσι ώστε να είμαστε πιο σαφείς και αποτελεσματικοί. Αποφασίσαμε λοιπόν να αφήσουμε στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να ασχοληθεί με τα ιδιαίτερα στοιχεία. Όμως εμείς είπαμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά και όχι μόνο για την ίδια την αγορά αλλά και για να πέσουν ε, οι τιμές τιμές προ όφελο των καταναλωτών. Εκεί βάλαμε και κάποια ειδικά στοιχεία όσον αφορά τους καταναλωτές. Ας πούμε, ε, ότι οι ποινές θα πρέπει να καθορίζονται βάσει της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές. Επίσης ε, θελήσαμε να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος ε, πρόκειται ε, και είπαμε μαζί και με τους συναδέλφους σκιώδης συγητές ότι θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και κατηγορηματικοί όσον αφορά τους κανονισμούς που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται προς όφελος των καταναλωτών. Δεύτερον, Είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να προοδεύσουν τα πράγματα, ε, κυρίως όσον αφορά τις... Ε, ε, assigned uh, between three institutions, the Commission, the Council and the European Parliament, which actually strengthens our hand. Το μνημόνιο συνεννόησης, καθώς επίσης και τις... Ε, κα... This is not as if a nuclear option that we are only asked at the end of... Και τις υπόλοιπες πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν κατά αυτή την έννοια να υπάρχει ε, συνεννόηση έτσι ώστε ο, ο στόχος να επιτευχθεί. Τρίτον, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε σαφέστερη άποψη όσον αφορά τις ε, κυρώσεις. Έχουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες επ' αυτού, γιατί θελήσαμε να αποφύγουμε μια κατάσταση ε, κατά την οποία ε, κάποιοι οικονομικοί, κάποιοι ενεργόντες στην αγορά να αποφασίσουν να εγκατασταθούν σε μια χώρα, γιατί εκεί μπορούν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση και λιγότερες κυρώσεις από ότι σε κάποια κάποια άλλη χώρα. Προετοιμάσαμε έξι ε, συμβαστικές τροπολογίες. όπου συμπεριλήφθησαν τα περισσότερα σημαντικότερα για τους περισσότερους συναδέλφους στοιχεία. Και για μία ακόμα φορά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την εξαίρετη συνεργασία, ε, τους σκιώδεις εισηγητές και να πω βεβαίως ότι εμείς ε, συζητήσαμε πάρα πολύ και με την ε, Επιτροπή Ήτρε που είναι αρμόδια επί της ε, ουσίας και πιστεύω ότι κάναμε τελικά καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρθρο 1, παράγραφος 1, τροπολογία 40, τέρμες. Υπέρ. Κατά. Τώρα ψηφίσαμε. Το ΕΛΚ δεν ψήφισε. Για να επαναλάβουμε. Τροπολογία 40. Είναι υπέρ κατά αποχές. Μάλλον, μάλλον απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε, παρακαλώ. We check amendment 40. We, we close. Α, απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 41. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Αρθρο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Amendment 42, 43. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, εντάξει. Δεν είμαι κι εγώ η ίδια πολύ σίγουρη. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεχίζουμε τροπολογία 12 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 4, τροπολογία 45 του κυρίου Μάντερς, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 45. πέρα στις ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ 16 κατά. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές. We will check it μάλλον να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Ε, ναι, 28 ψηφίσαντες, 28 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνο, ομόφωνο, μπράβο. Τι να σας πω, η πρόεδρος σας προφανώς δεν βλέπει καλά, λέει η πρόεδρος. Επόμενη τροπολογία του κυρίου Τόρνς υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εδώ πράγματι πρέπει να ε, ελέγξουμε. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Όχι, όχι, αυτή δεν ψηφίζεται. Θα πάμε απευθεία στην 52. 52 του εισηγητού και λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 15 απεσύρθη. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μάλλον όχι. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 49. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με διαφορά μίας ψήφου. 14 υπέρ 13 κατά δύο αποχές. Τροπολογία υπαριθμών 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7, τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 8, τροπολογία 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Φτάνουμε τώρα στο άρθρο 9, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε απευθείας λοιπόν στην τροπολογία 56, υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 13 ε, και συμβασική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση ή όχι. Όχι, όχι, δεν ελέγχουμε. Τροπολογία 15, 21 ε, στο άρθρο 15. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Άρθρο 16, τροπολογία 61. Απερίφθη ή ενεκρίθη. Η 21 να ελέγξουμε την τροπολογία 21. 21 λέει η Πρόεδρος. Πέρασε της ψηφοφορίας. Ναι, ναι, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Πού είμαστε τώρα. Τροπολογία 61. Παρακαλώ. Τροπολογία 61. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. And uh, we go to recitals Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην τροπολογία 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί, πηγαίνουμε στην τροπολογία 29. Εκεί έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Όχι. Εντάξει, συμφωνείτε ότι ε, ε, δεν έγινε αποδεκτή. Πολύ ωραία. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 31 με προσθήκη προφορικής τροπολογίας. So oral amendment replaces Προφορική τροπολογία ε, για να αντικατασταθεί το various European agencies με the agency υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34, επί σκέψη 15, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ελέγξουμε. η Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 37, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντως. Σαφώς, τέσσερις ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε συνάδελφε. Συνεχίζουμε λοιπόν τη μέσα διάταξη και φτάνουμε στο σημείο 6, έλεγχος των μεγάλων κινδύνων που συνδέονται με τα μείζων ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνε ουσίες. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάντσλικ, τη συντάκτρια της γνωμοδότησης. Παρακαλώ κυρία Χάντσλικ. Please, Mrs. Hanslick. Okay. Uh, colleagues, sorry. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να μιλήσω κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η οδηγία σε βέσο είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων. Απαιτούνται αλλαγές στην οδηγία. Συγκεκριμένα θέλουμε να υπάρξει τροποποίηση 1 στην ταξινόμηση, στην επισήμανση και στην συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ευκταία. Έχουν υλοποιηθεί αρκετές διατάξεις, συμφωνώ με αυτές και συγκεκριμένα τις διατάξεις οι οποίες αφορούν την πρόσβαση των πολιτών για την εισαγωγή των ε, διατάξεων προσφυγή στη δικαιοσύνη αναφορά ατυχημάτων. Η απλούστευση της αναφοράς, υποβολή των εκθέσεων ε, και τη ενημέρωση τη πληροφόρηση είναι κάτι πολύ θετικό. Στην έκθεση μου προτείνω κάποιε αλλαγέ. Οι αλλαγέ αυτέ αφορούν δύο στοιχεία. Το πρώτο ε, είναι το παράρτημα 1 το οποίο αλλάζει και δεύτερον ενημέρωση των, ε, του κοινού. Προτείνει η Κομισιόν κάποιες αλλαγές ε, στο παράρτημα 1 στο attachment 1, σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξης, κατάργηση κάποιων ουσιών και εισαγωγή κάποιων νέων ουσιών. Περί αυτού πρόκειται. Το attachment 1, το προσάρτημα 1, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οδηγίας γιατί ορίζει τις ουσίες και κάποιες οριακές τιμές. Ταυτόχρονα εξηγεί το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, τον αριθμό φορέων με βάση απαιτήσει της οδηγίας Ευρέσο 2. Νομίζω ότι αλλαγέ σε αυτό το παράρτημα, αλλά και στο παράρτημα 7, το οποίο περιλαμβάνει τις ε, παρεκκλήσεις από τα πρότυπα δυνάμει του άρθρου 4, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ενταχθούν ε, στην κανονική νομοθετική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο του παραρτήματος 1, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή μας υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι θέλησαν συμπερίληψη ή αφαίρεση κάποιων ουσιών. Αν δει κανεί το περιεχόμενο του παραρτήματος 1, Νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Δυστυχώς όμως ούτε εγώ ούτε η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχουμε την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για να ορίσουμε κατά πόσο μια συγκεκριμένη ουσία πρέπει να συμπεριληφθεί ή να μην συμπεριληφθεί στις ουσίες που απαριθμώνται στον κατάλογο του παραρτήματος 1. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση που έχω να σας κάνω αφορά μόνο τη διαδικασία της αλλαγής και όχι τις ίδιες τις ουσίες αυτές καθ' αυτές. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημοσιοποίηση των πληροφοριών, νομίζω ότι πέραν του καθήκοντος δημοσιοποίησης, είναι σημαντικό η ποιότητα και η μορφή της πληροφορίας να οριστεί με το σωστό τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένη πληροφορία, εύληπτη, εύκολα κατανοητή από τον πολίτη, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με τη συμπεριφορά των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όταν υπάρξει κάποιο σοβαρό περιστατικό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν οι σωστέ πληροφορίε. Η ποσότητα δεν είναι το σημαντικό, η ποσότητα των πληροφοριών, αλλά η ποιότητα. Να είναι δηλαδή ε, οι σωστέ πληροφορίε αυτέ που θα λάβουν οι πολίτες. Κυρίως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλοι δημόσιοι χώροι. Συμφωνώ επίσης με την πρόταση της Κομισιόν να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού με πιο ανοιχτό τρόπο θα έλεγα. Υπάρχουν βέβαια κάποια στοιχεία εμπιστευτικότητας. Υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οπότε οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται μόνο κατόπιν ετήματος. Κάθε τέσσερα χρόνια επίσης η Κομισιόν πρέπει να παρουσιάζει μια έκθεση σε σχέση με μείζωνα ατυχήματα ή ε, περιστατικά έκτακτης ανάγκης που συνέβησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να σχολιάζει, δηλαδή ποιος ήταν ο αντίκτυπος αυτών των ατυχημάτων ή αυτών των περιστατικών ε, και για τη λειτουργία της οδηγίας. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες θα ήταν πολύ χρήσιμες και θα έπρεπε να υπάρξει και περαιτέρω συζήτηση για την οδηγία σε ΒΕΣΟ 2. Αυτές είναι οι πληροφορίες, αυτά είναι τα σχόλια που έχω να κάνω για την οδηγία αυτή. 21 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι λίγη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα τον Ιούλιο. Τώρα θα ήθελα να ακούσω βέβαια με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή τα δικά σας σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι, συγγυ... οι Η κυρία Ίσμερ Μαρία Πέρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο και για το έγγραφο το οποίο μας έχει παρουσιάσει. Συμφώνω μαζί της ότι σκόπιμο θα ήταν η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή να είναι η Επιτροπή ΕΜΠΗ, αυτή που θα διατυπώσει την αρχική πρόταση. Αυτό σε ό,τι τη διαδικασία. Και όταν είχαμε ανταλλαγή απόψεων τον Απρίλιο με την εισηγήτρια, Είχαμε πει ότι η τροποποίηση του παρατήματο 1 δεν θα πρέπει να γίνει μέσω του μηχανισμού κατά εξουσιοδότηση πράξεων, όπω προβλέπει η Κομισιόν τροποποίηση αυτού του Παρατήματο που είναι σπονδυλική στήλη, σκελετός ε, της οδηγίας γιατί περιλαμβάνει τον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών ε, και τα κατώτατα όρια θα πρέπει να τροποποιείται μέσω τη κανονική, τη τακτική νομοθετική διαδικασία. Επίση συμφωνώ ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση είναι πολύ σημαντική. Οι πολίτες και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι ενδέχεται να πληγούν από σοβαρό ατύχημα, ιδίω όταν ένα ατύχημα έχει δυσνοριακές επιπτώσεις, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, μονίμως και διαφανώς στις απαραίτητες πληροφορίες. Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς επίσης και μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών για την πρόληψη αυτών των διασυνοριακών ατυχημάτων. Και τονίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία οι πληροφορίες που θα περιέχουν τα συστήματα που θα δημιουργηθούν για τα μεγάλα ατυχήματα να ενημερώνονται, να επικαιροποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να εκπονεί έκθεση κομισιών για τα σοβαρά ατυχήματα που, ε, θα, που θα έχουν λάβει χώρα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα τη οδηγία. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την περιοδικότητα των εκθέσεων, έχω κάποιε αμφιβολίε. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να εκπονεί τέτοιε εκθέσει κάθε φορά που υπάρχει ένα σοβαρό ατύχημα και ιδίω όταν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Έτσι θα μπορούμε να αξιολογούμε τι πληροφορίε που διαβιβάζουν τα κράτη-μέλη και να διατυπώνουμε και συστάσεις που θα επιτρέψουν να προλαμβάνονται ε, αντίστοιχα ατυχήματα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την εισηγητρία για την εξαιρετική της λέει και θα πω ότι και η ομάδα μας ε, θα καταθέσει τροπολογίες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρότσμαν από την άλλη είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος ε, της ε, αρμοδίας συναδέλφου που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό. Η κυρία Παρανόβα θα ήθελε να συγχαρεί ε, την εισηγήτρια για τις προτάσεις της και τις προτινόμενες τροπολογίες. η πρόθεση τροποποίησης των ε, παραρτημάτων 2 και 7 ε, μέσω κατεξουσιοδότησης ε, πράξεων βρίσκει σύμφωνη την συνάδελφό μου. Επίσης, η πρόταση για μείωση των οριακών τιμών και των κατοφλίων την βρίσκει σύμφωνη αλλά σημειώνει ότι ίσως δεν είναι σωστή η συστολή της, ε, του εύρους του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Όσον αφορά τις ουσίες μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά τις οριακές τιμές. Για ορισμένες ε, ε, ουσίες δεν είναι σαφής η επιστημονική αιτιολόγηση των αναφερομένων τιμών Ας πούμε, για τις διοξίνες ε, οι τιμές ε, κατοφλίων δεν εξηγούνται ε, επιστημονικά. Επίσης ε, ε, τα στοιχεία αυτά ε, είναι καλό που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 γιατί καταδεικνύουν την σημασία για την ανθρώπινη υγεία. Δεν μπορεί εκεί να μπουν ουσίες οι οποίες δεν είναι τοξικές. Η κυρία Παρανόβα ενδεχομένως θα ήθελε να προχωρήσει λίγο περισσότερο όσον αφορά την αναφορά μεγάλων ατυχημάτων. Στην πρότασή της θεωρεί ότι θα πρέπει να αναφερθούν περισσότερες ουσίες οι οποίες προκαλούν ε, ατυχήματα. Και επίσης ε, θεωρεί η κυρία Παρανόβα ότι θα πρέπει να γίνεται καλύτερη αναφορά ε, στους τοξικούς κινδύνους και θα πρέπει επίσης να αναφέρονται λεπτομερέστερα οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ότι θα πρέπει λεπτομερέστερα να αναφέρονται όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στο περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ που μιλήσατε εξ ονόμα της κυρίας Παρανόβα. Η κυρία Ρούλ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Βεβαίω το θέμα είναι αρμοδιότητες τη Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά πολύ ορθώς η συντάκτρια της γνωμοδότηση, κυρία Χάντσλικ, κρατήθηκε στα σημεία τα οποία ενδιαφέρουν τη δικιά μας Επιτροπή. Ε, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, δικαίωμα ενημέρωση, ε, οτιδήποτε δηλαδή αφορά την προστασία των καταναλωτών. Αυτό την ε, απασχόλησε περισσότερο και αυτό είναι καλό. Όσον αφορά τώρα τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, όλες τις συνήθεις νομιθετικές διαδικασίε, εδώ έχει βάλει ένα ερωτηματικό. Εγώ όμω πιστεύω ότι εδώ δίνονται πολύ θετικά στοιχεία βελτίωση της πρόταση τη επιτροπή. Επομένω περιμένω να ακούσω την άποψη τη Επιτροπή εάν και κατά πόσον μπορεί να δεχτεί τις ε, σωστέ αυτέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούλε. Μήπω η Γκούε μέσω κάποιου εκπροσώπου τη θέλει να πει κάτι, θέλει να σχολιάσει, γιατί δεν βλέπω τον σκιώδη εισηγητή εδώ. Οπότε στρεφόμαστε στην Επιτροπή. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, καλοδεχόμαστε το ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή σας στην πρότασή μας. Ε, φυσικά πρόκειται για μια οδηγία που έχει να κάνει με την προστασία και την ασφάλεια των προσώπων και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό βέβαια. Η αναθεώρηση της οδηγίας προκλήθηκε κατά βάση από αλλαγές ε, στην ε, ταξινόμηση των χημικών ουσιών που έχει εγκριθεί διεθνώς και πρέπει να ενταχθεί στην κοινωτική νομοθεσία. Άρα η οδηγία αυτή που αφορά την νομοθεσία των χημικών ουσιών πρέπει να ε, μπορεί να λειτουργήσει και μετά την αλλαγή του συστήματος χημικών ουσιών που θα γίνει το 2015 συμφωνούμε με την έμφαση που δίνεται από την εισηγήτριά σας αλλά και από τους διάφορους και που σήμερα μίλησαν, η σημασία λοιπόν που δίνεται στην πρόσβαση στην ενημέρωση. Για να υπάρχει πρόληψη επιτυχημένη και ε, αντιμετώπιση επιτυχημένη των ατυχημάτων θα πρέπει να υπάρχει ε, πολύ καλή ενημέρωση ε, του κόσμου για το ατύχημα, για τη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάζονται πάνω σε αυτήν την έκθεση που στηρίζουν τη διάταξη αυτή της πρότασής μας. Και βέβαια ότι θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες, μέρος τουλάχιστον της πληροφόρησης, στο διαδίκτυο, online. Αν δηλαδή κάποιος ε, είναι ε, θύμα ίσως κάποιο ατυχήματος, ε, θα πρέπει να ε, έχει άμεσα, γρήγορα πρόσβαση, γιατί μπορεί να είχε κάποιες πληροφορίες να τις ξέχασε, να τις έχασε. Θα πρέπει λοιπόν να διατίθενται στο διαδίκτυο. Και κατέουπιν πινετήματο πιο λεπτομερικές πληροφορίες να μπορούν να διατεθούν επίσης. Αλλά νομίζω ότι το θέμα αυτό των πληροφοριών που θα διατίθεται στο διαδίκτυο είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτά που είπε και η είναι πολύ σημαντικά. σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, σε ό,τι αφορά τι κατεξουσιοδότηση πράξης, θα ήθελα ε, να μου δώσετε ένα λεπτό για να σας εξηγήσω τι προσέγγιση προτείνουμε εμεί. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του όλου συστήματος. Έχουμε την κοινοτική νομοθεσία για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών. Κατά βάση χρησιμοποιούνται οι ε, διαθέσιμες πληροφορίε για τα ε, στοιχεία, για τις ιδιότητες των χημικών ουσιών για την ταξινόμηση αυτή. Όταν μια ουσία έχει ταξινομηθεί, δυνάμει της ομοθεσίας αυτής, εάν ε, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τοξικό παραδείγματο χάρη, ε, θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό υπόψη για την εφαρμογή τη οδηγία σε βέσο. Και βασιζόμαστε γι' αυτό σε τεχνικέ πληροφορίε. Και έχουμε τη ρυθμιστική διαδικασία με ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο βάσει και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτή είναι η συνήθι διαδικασία. Που από ό,τι ε, φαίνεται θα πρέπει να μεταφερθεί, να τροποποιηθεί και να ισχύει πλέον ε, πράξη οι ουσίες ταξινομούνται λόγω κάποιων εγγενών τους ιδιωτήτων. Αλλά ίσως αυτό να μην αντικατοπτρίζει το κίνδυνο, το βασικό κίνδυνο ατυχήματο. σε σχέση με τις συνθήκες χρήσης της ουσίας. Αν δείτε το τμήμα 3 του παραρτήματος 1, θα δείτε ότι δεν μιλάμε για αποκλεισμό μιας ουσίας από την οδηγία. Μιλάμε για καθορισμό των συνθήκων από τις οποίες μια ουσία εμπίπτει στην οδηγία ή δεν εμπίπτει στην οδηγία. Υπάρχουν πολύ καλώς καθορισμένα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει μείζον κίνδυνο ατυχήματο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί πάνω σε αυτό το σημείο. Αν χρησιμοποιούνται απλά ε, οι εγγενείς ιδιότητες, ίσως τελικά προκύψουν κάποια καταστάσεις επιταξινόμηση εγγενών ιδιωτήτων μέσω ε, της επιτροπολογίας να έχει έναν αντίκτυπο που δεν είναι ανάλογος ε, με τη σημασία ή την, το ενδεχόμενο υπάρξει ένα μείζον το θέμα είναι πώ ασκεί η ε, Κομισιόν τη εξουσία τη μέσω κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Εμεί έχουμε προτείνει το παράρτημα 4 που περιλαμβάνει κάποια βασικά, κάποια γενικά κριτήρια στα οποία θα πρέπει να βασίζονται οι αποφάσει. Και τώρα συνεργαζόμαστε με του εμπειρογνώμονε για να επαναπροσδιορίσουμε καλύτερα τα κριτήρια αυτά. Εν και του παραρτήματο 7 που θέλουμε να συμπληρώσουμε. Επίσης έχουμε εξετάσει και κάποια άλλα έγγραφα του Κοινοβουλίου που πιο πολύ έχουν να κάνουν με τα κριτήρια άσκησης των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων και όχι τόσο με την αμφισβήτηση του προσδιορισμού των κριτηρίων για το πώς θα ταξινομούνται οι ουσίες, αν θα εμπίπτουν ε, στην οδηγία σε βέσο και αν αυτά γίνεται μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων ε, προβλέπει η εισηγήτρια. κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αν πρόκειται για λιγότερο σοβαρά ατυχήματα θα μπορούσαμε μέσω των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί και των βέλτιστων πρακτικών να προχωρούμε. Υπάρχει μια πρόταση για μια επιπλέον έκθεση σε, επιπλέον σε σχέση με αυτή που προτείνουμε εμείς. Στο άρθρο 20, παράγραφο 4, λέμε ότι η Κομισιόν εκπονεί έκθεση, άρα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι η πρόθεση της εισηγήτριας να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή και να δημιουργηθεί ένας δεύτερος κύκλος υποβολής εκθέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ε, δύσκολο γιατί θα μας επιβαρύνει. Ήδη προτείνουμε και προβλέπουμε ένα κύκλο υποβολής εκθέσεων. Είπατε επίσης να υπάρχει έκθεση αμέσως μετά ε, κάθε ατύχημα. Κάποια ατυχήματα είναι πολύ μεγάλη εμβέλεια. Κάποια είναι σημαντικά, είναι μείζων ατυχήματα, αλλά έχουν περιορισμένες επιπτώσεις, περιορισμένο αντίκτυπο. Έχουμε 20 με 35 περίπου ε, ατυχήματα για τα οποία υποβάλλεται έκθεση κάθε χρόνο. Νομίζουμε ότι μετά από κάποια χρόνια, όταν θα έχουμε συγκεντρώσει ε, την επαρκή εμπειρία, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε στοιχεία για τα μείζωνα ατυχήματα και για την υλοποίηση της οδηγίας στην έκθεσή μας. Αλλά όχι να έχουμε έκθεση αυτή τη στιγμή τώρα ε, μετά από κάθε ατύχημα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Χάνσλι, μήπως θέλει να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την τόσο πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε πάνω στην εκθεσή μου. Έχοντας ακούσει τις ε, παρατηρήσεις σας, από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε σε μεγάλο ποσοστό κοινέ θέσει. Θα καταλήξουμε λοιπόν σε μια πολύ καλή συμβαστική λύση. Είναι καλό δείγμα αυτό για τον πρόοδο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι 21 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, λίγη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω το χρονοδιάγραμμα. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει 11 Ιουλίου. Ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ 12 Ιουλίου. Και στην Επιστουσία Αρμόδια Επιτροπή Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, που γίνει η ένβη αυτή και στην Ολομένα θα περάσει το Δεκέμβριο. Uh, here, so we... Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο 7. Για που είναι πολύ στην κυρία Γκέπχαρ. Τεχνικέ απαιτήσει για τι μεταφορέ πίσω και τι άμεσε χρεώσει ευρώ με την τροποποίηση του κανονισμού 924 2009. Θα με δώσω το λόγο κατευθείαν στην εισηγήτρια. Την κυρία Ευελίν Γκέφαρντ. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και πρόκειται για το θέμα της οργάνωσης του συστήματος ΕΠΑ και πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί και να οργανωθεί και διαμεθοριακά και σε κράτη-μέλη. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι προτάσεις που υπάρχουν, ε, που δεν δέχτηκε η Επιτροπή, θα μπορούσαμε να τις δεχθούμε. Δηλαδή να πούμε ότι θα πρέπει εκ παραλίλου να ε, λειτουργούν και τα παλιά συστήματα και το σύστημα ΣΕΠΑ. Πώς σκέφτηκα αυτό αλλά μετά ε, αναρωτήθηκα πώς θα δώσει μια τελική ημερομηνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σε μια εσωτερική αγορά που θέλουμε εμείς και σε ένα χρόνο ευρώ όπως τον θέλουμε δεν μπορούμε να έχουμε πολλαπλά συστήματα μεταφοράς πιστώσεων αλλά θα πρέπει να έχουμε κάτι πιο ενιαίο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αναρμόσουμε τα συστήματα. Äh, το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι τα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να ε, ζητήσουμε τη μεταφορά στο σύστημα ΣΕΠΑ. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις και στην κοινή γνώμη, σε εκείνους που προστατεύουν τους καταναλωτές και μεταξύ άλλων επίσης και για το θέμα καταρχήν κατά πόσο θα πρέπει να ορίσουμε την ίδια ημερομηνία για τη μεταφορά πιστώσεων και τις άλλες ε, υπηρεσίες πληρωμών. Είχα προετοιμαστεί στα αγγλικά και δεν θυμάμαι τους γερμανικούς όρους, συγγνώμη. Λοιπόν, αν θα πρέπει και για τη μεταφορά πιστώσεων και για την ε, ε, ανάληψη. Εγώ στην αρχή είχα πει θα είναι η ίδια ημερομηνία. Μετά όμως το ξανασκέφτηκα. Και νομίζω ότι τα δύο αυτά συστήματα είναι διαφορετικά. Και η αναγκαιότητα της προστασίας των καταναλωτών είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική. Στην ε, μεταφορά πιστώσεων νομίζω ότι είναι πιο εύκολο. Γιατί ο καθένας ορίζει την, ε, τα στοιχεία πάνω στην, ε, στο έγγραφο μεταφοράς και επίσης αυτά τα στοιχεία δεν μεταφέρονται στον παραλήπτη. Ε, είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα όμως με τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων. Δηλαδή, στην περίπτωση στην οποία δίνει κανένας μία μόνιμη εντολή σε μία τράπεζα να μεταφέρει κάποια χρήματα. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το θέμα αυτό μπορεί να τύχει και καταχρηστικής ε, μεταχείρισης. Και είχα επαφέ με τράπεζε που μου είπαν πραγματικά κάποια πρέπει να, πράγματα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα συστήματα ασφάλειας. Και η Κομισιόν προβλέπει διαφορετικές ε, καταληκτικές ημερομηνίες για την θέση εφαρμογή, δηλαδή για το θέμα των πιστώσεων είναι πιο σύντομο. και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προστατευτούμε για την άλλη τη μόνιμη μεταφορά από καταχρήσεις στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που έπρεπε να εξετάσουμε κατ' ουσίαν, όπου πρέπει να βρεθεί μια λύση από σκοπιάς προστασίας του καταναλωτή. Μετά, τι, πώς θα εξετάσουμε τις προθεσμίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκέφτηκα για μακρόν και το αυτό το θέμα. Και εν ώψη του ότι λέω ναι, να έχουμε μια, ένα ενιαίο χαρακτήρα των συστημάτων. Από την άλλη μεριά οι καταναλωτές θα πρέπει να συνηθίσουν και το καινούριο σύστημα θα πρέπει να προβλέψουμε νομίζω δύο χρόνια περισσότερα από εκείνα που προβλέπει η Κομισιόν. Δηλαδή τέσσερα χρόνια για την μεταφορά και πέντε χρόνια αντί τρία για την άλλη πράξη. Αυτό θα ήταν νομίζω λογικό, ούτω ώστε να μπορούμε να φροντίσουμε, να συνηθίσουν οι καταναλωτές αυτό το καινούριο σύστημα. Αυτό ήταν το, το δικό μου κίνητρο για την πρόταση μιας παράτασης των προθεσμιών έναντι αυτού που προτείνει η Εκτελεστική Επιτροπή. Αυτό βέβαια θα έχει και επιπτώσεις όσον αφορά την υποχρέωση παρουσίασης ε, έκθεσης από την Κομισιόν. Ε, γιατί βέβαια δεν περιμένουμε να υπάρχουν εκθέσεις εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του νέου συστήματος. Επίσης θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα παράδειγμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τα στοιχεία του οποίου εγώ συμπεριέλαβα στα εν λόγω άρθρα, γιατί πρόκειται για πολύ λεπτά θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Θα σας πω και ποια είναι η σχετική μου τροπολογία. Γιατί ίσως απορρίσατε βλέποντας ότι πρόκειται για μια πάρα πάρα πολύ μακρά τροπολογία. Αλλά είναι τόσο ε, Μα έχει γίνει τόσο μακρύ το κείμενο αυτό γιατί συμπεριλήφθησαν πολλά από τα στοιχεία του παραρτήματος όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσει για τις μεταφορές αυτές ε, πιστώσεων, ε, τη χρήση των ε, στοιχείων αυτών, τη μεταφορά των πράξεων πληρωμής, ανακοινώσεις. Λοιπόν, τόσο πάντων είναι πολλά τεχνικά θέματα ε, με τα οποία εμπλέκονται όμως και πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν τα άτομα εκάστοτε. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το εξαφανίσουμε σε ένα παράδειγμα που μπορεί να αλλάξει η Κομισιόν όπως θέλει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει στο κείμενο του κανονισμού γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τα οποία θα πρέπει και η πολιτική αρχή να έχει τη δυνατότητα επιβολής. Τροπολογία 26. ή μάλλον τροπολογία 31 που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και που ανέφερα ήδη. Πρόκειται το θέμα ποια είναι τα ρυθμιτικά στοιχεία που θα μπορεί να δει ο παραλήπτης όσον αφορά τον πληρωτή. Η Κομισιόν προτείνει και το όνομα του πληρωτή αλλά και ο αριθμός IBAN να αναφέρεται. Αυτό μου είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα, το οποίο δεν πρέπει απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία που δίνονται στον παραλήπτη. Αρκεί το όνομα. Έχει την ανάγκη και ο τόπος από τον οποίο αποστέλνω τα χρήματα. Αλλά το IBAN δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μεταβιβάζεται. Αυτή είναι επίσης μια πρόταση που κάνω. Ε, και υπάρχει και ένα τελευταίο στοιχείο. Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Και για τις επιστροφές αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το κόστος ποιο είναι το κόστος με το οποίο θα πρέπει να επιβαρυνθεί ο πληρωτής. Εγώ, με την τροπολογία μου υπαριθμών 12, προσπαθώ να διευκρινίσω τα πράγματα και λέω ότι ο πληρωτής δεν επιβαρύνεται για τις συναλλαγές τύπου Ε που προκύπτουν από ανεπαρκή ποσά στους λογαριασμούς του πληρωτή. Έως ότι η πληρωμή με άμεση χρέωση καταστεί απαιτητή. Και στο τροπολογία 13 λέει ότι εάν ο πληρωτής δεν είναι υπεύθυνο για τη ματέωση αυτών των συναλλαγών. Γιατί αν το πρόβλημα βρίσκεται στο τραπεζικό σύστημα, γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο πληρωτής. Όποιος ε, είναι υπεύθυνο για το κόστος αυτός, αυτό είναι εκείνος που θα πρέπει να επιβαρυνθεί. Νομίζω ότι αυτό συμπληρώνει πολύ καλά την πρόταση της Επιτροπής. Αυτά είναι τα σημεία που θα ήθελα να επιστρέψω τις σε αυτά και περιμένω να ακούσω με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις των συναδέλφων καθώς επίσης ε, και περιμένω με ενδιαφέρον να δω και τις τροπολογίες που θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο μέρες. Γι' αυτό και την περασμένη εβδομάδα όταν πήραμε τα μεταφρασμένα κείμενα αμέσως έστειλα το κείμενο αυτό στους ε, σκιώδεις ηγητές για να μπορέσουν να προετοιμαστούν έγκαιρα. Γιατί νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Και από την Επιτροπή ΙΜΚΟ να υπάρχει μια καλή γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΕΚΟ. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ κυρία Κέπχαρτ. Ο κύριος Μπουζούτιλ από το ΕΛΚ θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ κύριε Μπουζούτιλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Γκέπχαρτ για την ε, παρουσίαση της γνωμοδότησής της. Ε, θα ήθελα να περιστώ σε ένα σημείο που αφορά την προθεσμία αλλά όμως να ξεκινήσω λέγοντας ότι πράγματι πιστεύω ότι πρόκειται εδώ για πολύ σημαντική νομοθεσία όσον αφορά το συμφέρον ε, των ε, καταναλωτών και των επιχειρήσεων και αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε και την άποψη της ΙΜΚΟ στο νομοθέτημα αυτό. Το ζήτημα της ε, τελικής ημερομηνία είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ε, εισηγητής ε, της ΕΚΟΝ μας λέει ότι θα πρέπει να βάλουμε μία καταληκτική ημερομηνία μετά από μία διετία. Και πολλοί συμφωνούν ότι θα πρέπει αυτή η καταληκτική ημερομηνία να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη, γιατί θέλουμε να ολοκληρωθεί το σχέδιο αυτό γρήγορα και μία και καλή. Αυτή η ιδέα σέρνεται εδώ και πολύ καιρό και όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί, τόσο το καλύτερο και για τους καταναλωτές και για την εσωτερική αγορά και για τους ε, επιχειρηματίες. Η κυρία Κέπχαρτ, αν κατάλαβα καλά, θέλει να ε, επεκτείνει αυτήν την ημερομηνία από τα δύο χρόνια στα τρία χρόνια σε περίπτωση μεταφοράς πιστώσεων και στα τέσσερα χρόνια σε περίπτωση άμεσων χρεώσεων. Είμαι πεπισμένος όμως ότι δεν χρειάζεται μια τέτοια καθυστέρηση, ε, μια τέτοια επιμήκυνση. Από τα δύο χρόνια να πάμε στα τέσσερα είναι υπερβολικά μεγάλη επιμήκυνση. Ε, πραγματικά θα ήθελα να δώσω στην κυρία Γκέμπχαρτ όλο τον χρόνο που χρειάζεται ε, για να με πείσει ότι πρέπει να την στηρίξω σε αυτήν την ε, πρόταση επιμήκυνσης. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η φυσική μου τάση είναι να ακολουθήσω την πρόταση του επί της εισηγητού της επί επιτροπής γιατί πιστεύω ότι αυτό θα είναι προς όφελος των επιχειρηματιών, ε, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Αλλά πάντως ε, θέλω να με πείσει και η κυρία Κέπχαρτ, θέλω να μου πει τις απόψεις της για να με πείσει. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο ο κύριος Σολεσμίτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και βεβαίως ευχαριστώ και την συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Γκέπχαρτ. στην ουσία με κάλυψε ο κύριος Μπουζούτιλ. That's my Με κάλυψε λοιπόν ο συνάδελφος. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό, σημαντικότατο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις λοιπόν, αλλά και για τους καταναλωτές. Δεν πρέπει να σέρνουμε άλλο τα βήματά μας, Ίσως και εμένα μπορείτε να με πείσετε κάποια στιγμή, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω ότι θα αντισταθώ στεναρά. Δεν, δεν θα είναι εύκολο να με πείσετε, γιατί έχω μάλλον απεσιόδοξη στάση σχετικά με το κατά πόσο θα κερδίσουμε οτιδήποτε αναβάλλοντας ακόμα περισσότερο, επιμικίνοντας ακόμα περισσότερο την προθεσμία. Ελπίζω πάντως ότι θα πετύχουμε κάποια συμβαστική λύση στο τέλος. Κάτι άλλο. Ενδεχομένως θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες σχετικά με χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Και υπάρχει και το άρθρο 7.2. Δεν ξέρω αν η Γερμανίδα συνάδελφος θα το δεχτεί, αλλά πάντως εδώ πρόκειται για εξαίρεση η χώρα από την οποία προέρχομαι εξάγει κυρίως στη Γερμανία. Και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους καταναλωτές, ούτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε ειδικά καθεστώτα, ειδικέ ε, χώρες, εξαιρεσει κτλ. Αυτές είναι οι κύριες αντιρρήσεις μου, αλλά κυριότερο είναι το χρονοδιάγραμμα, κυριότερη αντίρρησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Äh, Κύριε Ρούλε, με συγχωρείτε. Ε, δεν είχα τη δυνατότητα να συζητήσω το θέμα με τον Πασκάλ Καφέ. Έχω όμω την εντύπωση ότι το θέμα του χρονοδιαγράμματο είναι ένα θέμα γερμανικό, αν θέλετε, η παράτηση αυτή που ζητιέται. Ε, τουλάχιστον έχουμε εκεί πολύ έντονη πίεση από την κοινή γνώμη. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ των πολιτικών και στο εσωτερικό της πολιτικής ομάδας. Εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω αν δεν έχω συνοηθεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους της ομάδας μου. Next speaker is from Γκουέ, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να πω πρώτα απ' όλα ότι προσπάθησα να πιστώ από το νέο χρονοδιάγραμμα αυτό, από το προτινόμενο παρατεταμένο ας πούμε χρονοδιάγραμμα σε, σε πολλές συνεδριάσεις, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να πιστώ, δεν βρίσκω ε, κανένα στοιχείο υπέρ ή επιχείρημα υπέρ της ε, και επομένως μάλλον θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μπουζούτιλ και τους άλλους συναδέλφους. Επίσης πιστεύω ότι δημιουργεί σύγχυση ε, και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και στους καταναλωτές. Πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, το ξέρουμε. Ενδεχομένως αυτό είναι δύσκολο για κάποιες χώρες, για κάποιες τράπεζες, αλλά δεν νομίζω ότι η δυσκολία είναι γενικευμένη και πιστεύω ότι υπάρχει σύγχυση που αυτή τη στιγμή υπάρχει το ευρωπαϊκό σύστημα και το εθνικό σύστημα και δεν ξέρουμε πότε θα χρησιμοποιήσουμε ποιο ή πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποιο και πώς θα γίνονται οι μεταφορές και πώς θα γίνονται οι χρεώσεις. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ε, στηρίζω την ε, ε, πρόταση της κυρίας Χάρτ. Επίσης, η ιδέα της να βοηθηθεί γενικότερα το κοινό και ε, όλα αυτά τα οποία αναφέρει, τα βρίσκω πάρα πολύ θετικά. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν και ένα αίτημα ε, βάσει του οποίου και εγώ υποβάλλω δύο τροπολογίες. Αυτή η ιδέα των καινοτόμων ε, συστημάτων πέρα από το διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, συστήματα τα οποία είναι καινοτόμα και καινούρια. Αυτό βεβαίως λέμε ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουμε οποιαδήποτε ε, καινοτομία ή εφαρμογή καινοτομίας ε, στον τομέα αυτό με τις προτάσεις μας βεβαίως δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή καινοτομίας ε, στον τομέα. και φυσικά να υπάρξει όλη η απαραίτητη εποπτεία του συστήματος. Αλλά κατά αυτή την έννοια είπα ότι θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στείλε. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτριά μας και θα ήθελα να μιλήσω για τις χρεώσεις. Οι τροπολογίες 12-13 της κυρίας Γκέπχαρτ είναι δεκτές και κυρίως η τροπολογία 15 στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ ε, που απευθύνει και η κυρία Γκέπχαρτ κάποιες ερωτήσεις ε, για την Κομισιόν σε σχέση με τις χρεώσεις. Εγώ είμαι από το Νομένο Βασίλειο, δεν είμαι βέβαια στην Ευρωζώνη, αλλά όταν έχω κάνει συναλλαγές μεταξύ Βελγίου ας πούμε και Νομένου Βασιλείου φαίνεται να υπάρχουν διαφορές από τη μια τράπεζα στην άλλη σε σχέση με τις χρεώσεις και όταν θα έχουμε ηλεκτρονικές ε, μεταφορές, ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτές τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο καταναλωτή όταν έχουμε ηλεκτρονική μεταφορά από μια χώρα στην άλλη, πάλι είναι δυσανάλογα υψηλέ αυτέ οι χρεώσει. Η ε, Επιτροπή Προστασία των Καταναλωτών υποτίθεται πρέπει να προστατεύσει του καταναλωτέ. Άρα είναι σημαντικό να κάνουμε αυτέ τι ερωτήσει δεν πρέπει να υπάρχει χρέωση για αυτού του είδους της πράξης, αυτού της συναλλαγής. Και αν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση, αυτό το τέλος θα πρέπει να είναι ισότιμο. Δηλαδή να ξέρει, ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, δυνατότητα καταναλωτές να γνωρίζουν ποιες είναι οι χρεώσεις από τη μια χώρα στην άλλη. Το θέμα των χρεώσεων νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τι έρευνα έχει κάνει η Κομισιόν ε, στα κράτη-μέλη, στις τράπεζες, σε σχέση με το κατά πόσον υπάρχει μία ε, χρέωση συγκεκριμένη ή αν υπάρχει τέλο πάντων προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Κύριε Κρότσμαν, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω θα πρέπει να το επιλύσουμε ευρωπαϊκά ή εθνικά. είναι η διαδικασία που έχουν οι τράπεζες για να τους αφαιρείται αυτόματα, λέγεται η πληρονή από τον, ε, ε, από τον λογαριασμό τους. Και πολλές τράπεζες ήρθαν επαφή μου και μου είπαν ότι ε, το κόστος θα ήταν τεράστιο για να αλλάξουμε το σύστημα και ο καθένας να εγκρίνει κάθε φορά. Και για να πούμε ας πούμε, ότι αν κάποιος έχει τόσο την έγκριση ήδη και αλλάξει το σύστημα, να μην χρειαστεί να ε, ε, κοινοποιηθεί στον καθένα ότι έχει αλλάξει ο αριθμός, γιατί τώρα έχουμε τον ευρωπαϊκό αριθμό και να πρέπει να εγκρίνει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά να γίνει αυτόματα αυτή η αλλαγή του αριθμού του δικαιούχου. Ε, αλλιώς θα κοστίσει εκατομμύρια, μου είπανε. Αυτό ισχύει για πολλά πράγματα, δηλαδή αποπληρωμή νερού, ηλεκτρικού, ε, συνδρομές, επιρροτικά κλπ. Θα υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία γιατί η σύμφωνη γνώμη για ένα νέο αριθμό ε, τράπεζας για τον ίδιο παραλήπτη δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Ιδίω αν παραμείνουν αυτέ οι πολύ σύντομε προθεσίε, θα πρέπει να το εγγράψουμε. Ξέρω, ξέρω το πρόβλημα τη προστασία των δεδομένων, κυρία Γκέπαρτ. Το καταλαβαίνω, αλλά ας πούμε οι, η οι λογαριασμοί τώρα είναι κάπως διαφορετικοί, δηλαδή είναι και ο παλιός αριθμός λογαριασμού μέσα σε αυτόν τον καινούριο ε, αριθμό ΣΕΠΑ, γιατί να μην το λύσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πούμε εντάξει, πρόκειται για μια τεχνική αλλαγή και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Γιατί κυρία Γκέπαρτ, καλό είναι να κάνει κανένας ε, να ακολουθεί αυτό το σύστημα. Εάν κανένας γράψει το λάθος ε, αριθμητικό στοιχείο, το έχω κάνει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Στη Γερμανία μπορώ να πω ότι όχι, έκανα λάθος, δεν χρειάζεται να πω γιατί και πώς και μου επιστρέφουν τα χρήματά μου. Ε, τουλάχιστον στη Γερμανία είναι έτσι το σύστημα. Γι' αυτό αν πάρουμε ιδίως τις σύνομες προθεσμίες να λύσουμε έτσι το πρόβλημα. Να το πούμε δηλαδή, να το θεωρήσουμε σαν μια τεχνική αλλαγή. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας αυτό γιατί ακριβώς σε εμά στη Γερμανία είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα γιατί μιλάμε για εκατομμύρια στοιχεία. Μήπως μπορούμε λοιπόν πραγματικά να το λύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και τα κράτη-μέλη μετά να έχουν κάποιες προθεσμίες μεταβατικές γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει και να ε, προσαρμοστούν οι τράπεζες. Αν το αφήσουμε το θέμα στο εθνικό επίπεδο, κύριε Πρόεδρε, θα έχει η τράπεζα περισσότερα προβλήματα. Θα πρέπει να περιμένει τι αλλαγή θα γίνει σε κάθε χώρα, αν θα είναι τεχνική, αν θα είναι ουσιαστική. Και γι' αυτό ας πούμε να προσπαθήσουμε να το λύσουμε έτσι αυτό το θέμα και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και πιο σύνομε ε, Ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Παρακαλώ. Α, όχι. Ναι, ναι, παρακαλώ κυρία Στέλλα. Ο κύριος ε, ε, Κρόιτσμαν αναφέρθηκε ε, σε κάτι που δεν ισχύει στη δικιά μας ε, χώρα. Ε, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτές οι πάγιες πληρωμές είναι άλλο πράγμα από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα εγώ. Μήπως μπορούμε να έχουμε και αυτή την αποσαφήνιση βεβαίως. Ναι, κάποια σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα σχετικά ε, με, το ίδιο, με την ίδια καταληκτική ημερομηνία που βεβαίως είναι και το πολιτικό ζήτημα αυτού του κανονισμού. Η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει δύο φιλόδοξες καταληκτικές ημερομηνίες, ε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2008 το πρόγραμμα για τις μεταφορές πίστοσης και ότι ήδη τον Νοέμβριο του 2009 ξεκίνησε αυτό για τις άμεσες χρεώσεις. Κάποιες ε, χώρες και κάποιοι ιδιωτικοί οργανισμοί ενδεχομένως έχουν ήδη μπει στο ΣΕΠΑ, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι ε, ε, ε, εμπορευόμενοι και κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί ακόμα. Άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν θα πρέπει να κυρωθούν τελικά, να υποστούν κυρώσεις τελικά αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη κάνει όλες τις προσπάθειες για να μπουν στο ΣΕΠΑ. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν κατά αυτήν την έννοια να δώσουμε, να, να αναφέρομαι μία φιλόδοξη καταληκτική ημερομηνία για την συμπερίληψη στο ΣΕΠΑ. Είπαμε λοιπόν ένα χρόνο για τις μεταφορές πίστοσης και δύο για τις ε, άμεσες ε, χρεώσεις. Έτσι ώστε να πιέσουμε όλους όσους δεν έχουν καν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μπουν στο ΣΕΠΑ να το κάνουν. Η κυρία Γκέμπχαρτ έκανε κάποιες ε, προτάσεις ε, μετακίνησης ή τροποποίησης ε, τμήματος του παραρτήματος στο κύριο σώμα των προτάσεων. Ε, εκεί όμως αναφέρονται πρόνοιες ε, οι οποίες αφορούν την προστασία των καταναλωτών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, τα νέα συστήματα γιατί η ΣΕΠΑ θα είναι η πρώτη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς πίστοσης ή άμεσης χρέωσης διασυνοριακά. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ε, προσθεθούν κάποιες επιπλέον πρόνοιες στους υπάρχοντες ε, κανόνες έτσι ώστε η μετάβαση να είναι πιο εύκολη, ε, η δυνατότητα επιπλέον ελέγχων να είναι επίσης πιο εύκολη ή εν πάση περιπτώσει να, να υπάρχει δυνατότητα περιορισμού ή άρνησης από πλευράς κάποιων μεταφορών πιστώσεων ή άμεσων χρεώσεων με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει επίσης και μία σειρά στοιχείων που θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρονται. Αυτά τα τεχνικά στοιχεία, εγώ πιστεύω, ε, και τεχνικά ε, χαρακτηριστικά θα πρέπει να παραμείνουν στο παράρτημα. Δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο σώμα της ε, οδηγίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί βεβαίως στην καινοτομία. Αυτό είναι ένα στοιχείο επί του οποίου συμφωνούμε. Θα πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι έτσι ώστε να συνεχίσει η δυνατότητα καινοτομίας και εξυγχρονισμού των τρόπων πληρωμών. Επιμένω, τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να μείνουν στο παράρτημα έτσι ώστε να ε, μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους ε, τροποποίηση των τεχνικών ε, χαρακτηριστικών. Όσον αφορά την καινοτομία, βεβαίως είναι σημείο κλειδί. Φυσικά δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε οποιαδήποτε χρήση της καινοτομίας. Παρ' όλα αυτά, οποτεδήποτε έχουμε πληρωμές ε, μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω ε, διαδικτύου. Όποτε υπάρχει μεταφορά πίστοσης ή άμεση χρέωση, ως μέρος του ε, τρόπου πληρωμής, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει αυτή η πληρωμή να εμπίπτει στο πεδίο της οδηγίας. και όποτε θέλουμε να κάνουμε πληρωμές με άλλο πιο διαφορετικό τρόπο, τότε σαφώς δεν εμπίπτουν σε αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστοσης και άμεσες χρεώσεις. Τέλος, σχετικά με τις χρεώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά μόνο το θέμα των χρεώσεων που, πληρών, που χρεώνονται μεταξύ, ε, μεταξύ τραπεζών. Και μπορεί να καθοριστούν διμερός ή πολυμερός. Η χρέωση του καταναλωτή καλύπτεται ήδη από υπάρχοντα κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές. Εκεί έχει τεθεί η αρχή της ίσης χρέωσης. Η ίδια χρέωση δηλαδή ε, για, για, για συνδιαλλαγές που αφορούν τη χώρα ή που αφορούν διακρατική ε, συναλλαγή. Εκεί θα πρέπει, λέμε, να είναι ίδιες οι χρεώσεις και αυτό δεν αλλάζει. Όσον αφορά δηλαδή τη χρέωση που τελικά χρεώνεται ο καταναλωτής. Και πρέπει να πω ότι ε, βάσει αυτής της αρχής είχαμε μια γενικευμένη μείωση των χρεώσεων που ε, έβαζαν οι τράπεζες ε, προς τους καταναλωτές. Δηλαδή μειώθηκε η δια, διασυνοριακή συναλλαγή στο ύψος της ε, εσωτερικής συναλλαγής. Εδώ, σε αυτήν τον κανονισμό, αναφερόμαστε στο πολυμερές ε, στοιχείο της, ε, των μεταφορών πιστώσεων ή άμεσων χρεώσεων βάσει των αρχών της υγιούς ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει γενικευμένη ε, απαγόρευση επιπλέον χρεώσεων για κάθε συνδιαλλαγή. Όμως ενδεχομένως ε, μπορεί να υπάρξει ένα πολυμερές σύστημα μονάχα για τις συναλλαγές αυτές ε, οι οποίες αφορούν επιστροφή χρημάτων ε, για μία από τις τράπεζες. Εδώ δεν αναφερόμαστε, ε, επαναλαμβάνω, στην χρέωση την οποία καλείται να καταβάλει τελικά ο καταναλωτής. Αυτά είναι τα σχόλια τα οποία ήθελα να κάνω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να ε, απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μια ομάδα ε, πολύ εξαχόντων καλεσμένων που θέλω να καλωσορίσω. Είναι γερουσιαστές από την ζυχία Θέλω να τους καλωσορίσω. Είναι προσκεκλημένη της κυρίας Ρόιτοβα. Καλώς ήρθατε. Speaker. Επόμενος ομιλητής, επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Γκέπχαρτ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτο σχόλιο. οι πρώτες μου παρατηρήσεις για τα τέλη αφορούν τις επιστροφές και όχι όλα τα άλλα τα οποία είχα αναφέρει στο παρελθόν. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει καμία αντίφαση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ μονάχα άλλαξα τη τάξη μεγέθους, γιατί αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ πολύπλοκο. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο απλοί. Άμα να το συστήσουμε πάντως. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω για πολλά πράγματα. Όπως είπε και ο κ. Τεζόν, δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τις καινοτομίες, δεν θέλουμε να έχουμε πολλές εξαιρέσεις. Κύριε Τεζό, ακριβώς προτείνω τη διαγραφή του άρθρου 7 γιατί προβλέπει πάρα πολλές εξαιρέσεις. Προσπάθησα επίσης να προβλέψω μια απλούστευση όσον αφορά την ε, παράταση ή μη παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή της, ε, ε, του κανονισμού αυτού. Εγώ για τις άμεσες πληρωμές δεν προ... παρατείνω από 2 σε 4, όχι, από 3 σε 4, δηλαδή κατά ένα έτος σχετικά με αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Ένα αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που με έκαναν να υποβάλω αυτή την πρόταση. Πρώτον, οι ομάδες προστασίας των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητούν να αφήσουμε ε, να λειτουργούν και τα δύο συστήματα, και το ΣΕΠΑ και το εθνικό χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Θα ήταν και αυτή μια δυνατότητα. Άλλοι νόση λένε να το κάνουμε αμέσω. Εγώ σκέφτηκα λοιπόν τώρα πού θα βρίσκαμε το συμβιβασμό ανάμεσα σε αυτές τις διάφορες θέσεις. Και όπως είπε και η κυρία Ρούλε, από δική μου χώρα, ξέρω όσον αφορά τις αρχές, τι τοπικέ αυτοδιοικήσεις παραδείγματος χάρη, φοβούνται ότι σε αυτά τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται δεν θα τα καταφέρουν. Και γι' αυτό σκέφτηκα ότι αν έχουμε μια παράταση αυτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν είναι και τόσο τραγικό. Γιατί συχνά πρόκειται για τα μικρές ε, κοινότητες που Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Υπάρχουν δυσκολίε με κάτι τέτοιο. Ένας είναι ο λόγος γιατί προτείνω μια παράταση κατά ενός έτος σε σχέση με αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί θεωρώ επίσης ότι κατά τα άλλα θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές ε, ε, ε καταλεκτικές ημερομηνίες για τον δύο ειδών της πληρωμές γιατί πιστεύω ότι είναι διαφορετικά τα συστήματα της πληρωμής και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποια διαφορά μεταξύ τους. Βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Γολτσμαν. Σημαντικό. Είχα κατά νου να υποβάλω μια τροπολογία. Τώρα δεν τη βρήκα εδώ στο κείμενο, σα ξέχασα να την υποβάλω. Αλλά είναι κάτι που μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλα αυτά. Γιατί εγώ θα ήθελα να υπάρχει μία διάταξη ότι για τις μόνιμες εντολές, για τις άμεσες πληρωμές που έχουν ήδη χορηγηθεί στην τράπεζα, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Εγώ τώρα άλλαξα την τράπεζα και ανάσκασα να τα κάνω, να κάνω όλες αυτές τις αλλαγές και ξέρω τι σημαίνει. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα χρειάζεται να αλλάξουμε, αλλά αυτόματα να γίνει αυτή η αλλαγή. Προσπάθησα να βρω την τροπολογία αυτή, που έκανα ή που νόμιζα ότι έκανα, αλλά δεν τη βρήκα. Ε, θα την ξαναυποβάλω. Αλλά και εσείς άμα θέλετε μπορείτε να την υποβάλλετε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θα πρέπει να γίνεται για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι αυτό επιλύει τα σημαντικότερα θέματα που εθίγησαν και τώρα περιμένουμε ανυπομονησία τις τροπολογίες και την συνεννόηση με τους κοιόδης ηγητές για να δούμε πως, πώς μπορούμε να πετύχουμε και ε, συμβιβασμούς για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ε, καταναλωτές, ε, τα στοιχεία των καταναλωτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ για τις αποσαφηνήσεις σας. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 25η Μαΐου τρέχοντος έτους στις 6 το απόγευμα. Και την 15η Ιουνίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες αυτές και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια πλέον, στην 1η του Σεπτεμβρίου. Όμως, να σας υπενθυμίσω ότι έχει ήδη δημοσιευθεί το νέο newsletter της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Και θα το βρείτε έξω από την αίθουσα, δίπλα στην είσοδο. Και βεβαίως ε, μπορείτε να γίνετε φίλος του newsletter και να το λαμβάνετε προσωπικός. Σημείο 8. Συμβάσεις πίστοσης για ακίνητα κατοικίας. Ο συντάκτης παρακαλώ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist jetzt Verbraucherkredit die zweite. Ich freue ε, χαίρομαι που βλέπω ορισμένους συναδέλφους εδώ που ήταν ήδη και στην πρώτη, πρώτη θα έλεγα, ε, έκδοση αυτού του κειμένου και τώρα έχουμε τη δεύτερη έκδοση. Χαίρομαι που αντέξατε τόσα χρόνια. Να σας πω στα λίγο να περί πρόκειται. Ε, για τις ε, υποθήκες δεν υπάρχει τίποτα μια που εξαιρούνται από την οδηγία για ε, τις πιστώσεις κατανάλωσης. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όμως αυτά αυτού του τύπου οι συμβάσεις πιστώσεων για τα τα υποθήκες δηλαδή. Και σας το λέω γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε εντάξει να μην επικαλύπτονται, αλλά να μην υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη και στην οδηγία για την, ε, υποθηκών για κίνητα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ καλό που η Κομισιόν δεν θέλησε να αλλάξει τα πάντα εδώ αλλά η πρότασή της είναι ευχάριστα σύντομη. Και εγώ θα ήθελα να πω αυτό που λέγει η Κομισιόν. Άλλο η καταναλωτική πίστη, άλλο η πιστώσεις για τα. Γιατί η καταναλωτική ε, πίστη είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την διακίνηση από τα σύνορα όταν αγοράζει κανένα με τηλεόραση ή ένα αυτοκίνητο και υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν ορισμένε ε, ρήτρες που δεν έχει υπόψη του ο καταναλωτής. Αλλά όμως η πίστοση για την ε, ε κατοικία, για το ακίνητο, πολλές φορές αναγκάζεται κανένας μας να πάει και στο συμβολιογράφο για να πάρει αυτό το τύπου το δάνειο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση παρεξηγήσεων. Και είναι και περιορισμένε δυνατότητες βέβαια ε, εσωμάτωση σε άλλες γιατί δεν υπάρχει το πρόβλημα γλώσσα, δεν υπάρχει το πρόβλημα της εμπιστοσύνη στην, ε, στην τράπεζα, αλλά υπάρχει και το θέμα της ε, ε της χρηματοδότησης ε, από την τράπεζα, μέσω μιας άλλη τράπεζα μέσω ενός οργανισμού που δεν γνωρίζει ο καταναλωτή. Αυτά είναι προβλήματα που παρεμποδίζουν μια πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς. Αλλά βέβαια δεν θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα πάντα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό πραγματικά και η Κομισιόν είναι πολύ επιφυλακτική. Καταρχήν, Τώρα, ε, παιδεία Οποιαδήποτε πίστοση ε, καλύπτεται με μια υποθήκη ή, ή μια πίστοση που πραγματοποιείται για την αγορά κατοικίας χωρίς να καλύπτεται από την υποθήκη. Και οι δύο περιπτώσεις καλύπτονται από ότι πρέπει να καλύπτω από την οδηγία τουλάχιστον. η οδηγία την κανονική πίστη προβλέπει εξαιρέσεις που δεν θα προβλεφθούν νομίζω. Θα σας τις αναπτύξω στην έκθεσή μου. Δεν είναι τόσο σημαντικό νομίζω. Απλώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ε, συνεπείς. Ένα πρόβλημα της οδηγίας αυτής είναι όταν ζητάτε ζητάτε να διαβάσετε ποια είναι η εμβέλεια οδηγίες, λέει οι εμβέλειες οδηγίες είναι συμβάσεις πιστώσεων. Αυτό όμως ε, είναι πολύ γενικό. Θα πρέπει να πούμε περί τίνος πρόκειται να μην ανατρέχουμε στους ορισμούς. Μήπως η Κομισιόν θα μπορούσε να διατυπώσει διαφορετικά να μας εξηγήσει γιατί το κάνει αυτό. Άρθρο 5. Λέει ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του καταναλωτή. Ε, ναι. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη βέβαια τα συμφέροντα του καταναλωτή, αλλά για το βέλτιστο συμφέρον δεν ξέρω αν δεν θα πρέπει να το επανεξετάσουμε είναι κάπως περιοριστικό αυτό μου φαίνεται. Ή μάλλον θα πρέπει να έχουμε εμείς μια πιο περιοριστική διατύπωση. Μετά όσον αφορά τις ικανότητες των υπαλλήλων των τραπεζών. Ναι, να έχουν κάποιες ικανότητες γνώσεις, αν έχουν υπερβολικά πολλές όμως θα είναι πολύ ακριβή, οπότε αυτό θα ακριβίνει την πίστοση. Οι πληροφορίες πριν από την υπογραφή της σύμβασης διακανονίζονται, αλλά δεν ξέρω, είναι θέμα της ε, τράπεζας να αναφέρεται στη δυνατότητα έκπτωσης ε, των ε, τόκων από τον ετήσιο φόρο του καταναλωτή. Μου φαίνεται υπερβολικό. Αυτά που είναι καλά και λογικά δεν θα πρέπει να συμπεριλάβονται απαραίτητο σε ένα νομοθετικό κείμενο ίσως ένα δελτίο πληροφόρησης να μπορεί να χορηγηθεί. Τέλος, κάποιες ε, εξηγήσεις που θα πρέπει να δοθούν και μετά ο πραγματικός ετήσιος τόκος. Ε, λέγεται ότι το κόστος της ασφάλειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο επιτόκιο αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι που διαφέρει από χώρα σε χώρα και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί. Εάν πρέπει να αναφέρεται και στην ε, διαφήμιση, αποκλείεται να αναφέρεται αυτό το ποσοστό του επιτοκίου, γιατί δεν είναι λόγω της ασφάλειας που πρέπει να συμπληρωθεί ξεκάθαρο. Μετά, την εφαρμογή. Θα πρέπει ίσως να επιλέξουμε την, την διατύπωση για την εφαρμογή που αναφέρεται στην οδηγία για την κατανολική πίστη όσον αφορά το αξιόπιστο του ενδιαφερομένου. Επίσης λέγεται ότι αν ο καταναλωτής διαφαίνεται σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τράπεζας ότι δεν θα μπορεί να επιστρέψει το δάνειο, τότε θα πρέπει να του αρνηθεί το δάνειο η τράπεζα. Αυτό το πρέπει όμως είναι υπερβολικά ε, περιοριστικό. Γιατί η τράπεζα, άμα θέλει, μπορεί να πει θα του δώσουμε το δάνειο και ας ε, ε, έχει την ευκαιρία αυτή ο άνθρωπος να δράσει. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των πληροφοριών που πρέπει να δώσει ο ενδιαφερόμενος ε, καταναλωτής, ότι θα πρέπει να υπάρχει το θέμα της ε, προστασίας των δεδομένων αυτών, ότι η, ε, οι συμβουλές που θα δοθούν στον ε, καταναλωτή θα πρέπει να δίνονται ανεξάρτητα από τη χορήγηση του δανείου και γι' αυτό θα πρέπει να κοστολογούνται ξεχωριστά, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ε, πολλές φορές συμπεριλάβονται στο κόστος του δανείου και αυτό δεν είναι σωστό. Μετά, τι γίνεται στην περίπτωση προώρης επιστροφής. Είναι μακρύ η συζήτηση αυτή. Αν ε, θέλετε να ικανοποιήσετε το μαζοχιστικό σας εγώ, να διαβάσετε τις λεπτομέρειες της ε, οδηγίας για την κατανοητική πίστη σχετικά με το θέμα αυτό. η διατύπωση που έχει επιλέξει η Κομισιόν μου φαίνεται ότι αξίζει πραγματικά να βρει την σύμφωνη γνώμη μας, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, πόσο ακριβείς ε, μπορούμε να είμαστε. Λέγεται, ας πούμε, δεν επιτρέπεται να παρεμποδιστεί υπερβολικά ε, πώς θα μπορούμε να ορίσουμε το ότι είναι το υπερβολικά, υπερβολική παρεμπόδιση. Επίσης αναφέρεται ποιο άρθρο είναι αυτό, 12. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει υπερβολικό κόστος. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει κόστος. Γιατί κόστος, ο, στα αγγλικά ας cost μπορεί να συμπεριληφθεί και το, ο τόκος που καταβάλλεται. Στο άρθρο 1 σε 1 αναφέρονται ρητά ή τόκοι, αλλά όσον αφορά την πρόορη επιστροφή, όσον αφορά το κόστος που πρέπει να συμπεριληφθεί, δεν αναφέρονται ε, καθόλου οι τόκοι. Ε, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τόκου στην πρόορη αυτή επιστροφή. γιατί αλλιώς υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και απειλείται και η πολυμορφία των προϊόντων που μπορούν να ε, έχουν πρόσβαση σε αυτά οι καταναλωτές. Αλλιώς δεν έχω τίποτα να πω όσον αφορά την πρώτη επιστροφή. Ίσως κάτι μπορούμε να συμπληρώσουμε στις διατυπώσεις σχετικές. Αυτά για τα συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, θα ήθελα γενικά να σας πω ότι ε, λέγεται κάπου ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν ξέρω, μπορούμε να το αφήσουμε έτσι και ολο... εν, ε, κατακλείδη υπάρχει εναρμόνιση λέγεται. Τι θα εναρμονιστεί ακριβώς και ποια, πότε. Αυτό δεν το λέει η οδηγία. Και μία ε, παρατήρηση, δηλαδή νομίζετε ότι αυτό θα γίνει έτσι αυτόματα ο τύπος παραδείγματος χάρη των εμπορισμών του πραγματικού φτώκου ότι θα ισχύει αυτό για όλα τα κρατημέλη και κανένα κράτος μόνος δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνει ή θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια λιγμό. Η θεωρειται οτι υπαρχουν λοιπόν, καποια περιθωρια λιγμου η είναι μια καλή βάση που χρειάζεται κάποιε διορθώσει, κάποιες διευκρινήσεις από δική μου σκοπιάς. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η κατεξοδιώτηση πράξη Χθε το συζητήσαμε με τον ε, Επίτροπο Μπανιέ στην ε, ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Εγώ είμαι υπέρ των κατεξοδίων συμπράξεων. Δεν θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πράττει σωστά όταν θέλει να ασχοληθεί με κάθε λεπτομέρεια. Αλλά αυτό ισχύει κυρίως για οδηγίες που αφορούν μηχανήματα και σκάλες, ε, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, αλλά δεν επιτρέπεται παντού και πάντα ε, να προβλέπει η Κομισιόν ε, πράξη, πράξης, παραδείγματος χάρη, τι είναι ο πραγματικός φτώκος, ε, τι είναι η παράταση των όρων δανειοδότησης κλπ. Αυτό είναι κάπως υπερβολικό νομίζω και δεν μπορούμε να το δεχτούμε όλα αυτά να γίνονται με κατεξιδότητες πράξεις. Ε, μετά δεν κατάλαβα γιατί οι προθεσμίες είναι τόσο σύντομες ε, που ορίζει η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, δεν είναι και τόσο τεράστια γιατί για αυτή ούτε θα αποτρέψει την οικονομική κρίση. Θα πρέπει να είχαμε περισσότερο καιρό στη διάθεσή μας. Αλλά εντάξει, αν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, αφού και η οδηγία δεν είναι και πολύ ογκώδης, ε, μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες αυτές. Εγώ θα ήθελα οι συνάλφοι κάτι να πούνε στα επιμέρους σημεία. Αλλά δεν θα πρέπει εμείς να διευρύνουμε την ευέλεια της οδηγίας αυτής, αλλά να παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια της πρότασης με διευκρινήσεις και με διορθώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And the next speaker... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόανκ Γκόγκ είναι ο επόμενος ομιλητής από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριε μάλλον Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς χαίρομαι που η Κομισιόν ε, ενισχύει τους όρους ε, για τις ε, πιστώσεις υποθηκών. Είναι μια πρακτική συνήθιση στα κράτη-μέλη. 6-3 ε, είναι το ποσό στην Ένωση και ο καταναλωτής δεσμεύεται για τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από 20 έως 30 χρόνια για αυτές τις ε, πιστώσεις και έχουμε και πολλές ε, αθετήσεις πληρωμών από νοικοκυριά που ξέρουμε και ότι αυτή ήταν και η αιτία της οικονομικής κρίσης η αδυναμία αποπληρωμή. Η κατάσταση όπως, σε χώρες όπως η Ισπανία δείχνει ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο επικίνδυνο που οδηγεί σε υπερχρέωση και σε προσωπικά οικογενειακά δράματα. Ε, μπορεί αυτό να οδηγήσει μέχρι και σε κατάσχεση της ε, περιουσίας και να ρίξει πραγματικά στο δρόμο τον ε, ε ανίκανο να πληρώσει το χρέος του πελάτη. Σε σχέση λοιπόν με αυτές τις ε, συμβάσεις πίστοσης, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι με ανησυχεί ένα θέμα διαδικαστικό. Υπάρχουν αρκετές πτυχές της πρότασης οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την προστασία των καταναλωτών. Τομέας αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής ΙΜΚΟ είναι αυτός. Όμως η αρμόδια καθήλυν ε, Επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε μια διαδικασία που θα εξασφαλίζει ότι το κείμενο της γνωμοδότησής μας θα ενταχθεί στο ακέραιο στην έκθεση Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα ήταν λυπηρό η γνωμοδότηση των μελών της Επιτροπής ΙΜΚΟ να μην ε, ληφθεί σοβαρά υπόψη, να είναι λίγο ε, αποδυναμωμένη όταν μιλάμε για θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Εγώ είμαι και μέλο Επιτροπή ΕΚΟΝ και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με βάση το άρθρο 51 στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Σε ό,τι αφορά τώρα την ίδια την πρόταση, θα περιοριστώ σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, τα συναφή προϊόντα, οι ε, συνδεδεμένα προϊόντα για την ε, αποδοχή της πίστοσης των τέτοιων ιατρινιών προϊόντων, μια υποθήκη που είναι ένα σημαντικό εχέγγυο, μπορεί κανείς να διερωτηθεί σε ποιο βαθμό παράπλευρες εγγύσεις, δηλαδή να ανοίξει λογαριασμό στο πιστοτικό έδωμα κτλ. Ο, ε, ο φιλέτης, μήπως αυτό οδηγήσει σε καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος του καταναλωτή. Δεύτερον, μια σημαντική πτυχή στη διάρκεια αυτής της περίοδου βλέπουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των, της αδυναμίας εξυπηρέτησης ε, αποπληρωμής ε, του, ε, της πίστοσης. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να υπάρχει προσφυγή υποχρεωτική σε διαιτησία και θα πρέπει επίσης να προβλέπω ότι αυτές τις πληρωμών λόγω ενός ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει ίσως σε ανικανότητα ή και σε πιο, να έχει πιο σοβαρές μοιρές συνέπειες και γενικά να, μπορεί να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να έχει στην αποπληρωμή του δανείου ο χρέο της. Αυτά είχα να πω και βέβαια θα ε, επαφηθώ και εγώ στην σοφία του εισηγητή, ο οποίο θα εμβαθύνει σε όλα αυτά τα θέματα. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Μπουσούα Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση μια σύμβαση ε, για την αγορά μια κατοικία. Και μπορεί ε, να κρατήσει ίσως και για όλη μας τη ζωή αυτή η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε οι καταναλωτέ να επιλέγουμε με τα γνώσεως. Μία πτυχή πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την πρόταση είναι ότι πρέπει να λαμβάνει πλήρεις ε, κατανοητές αντικειμενικές πληροφορίες από ευθύς εξ ο καταναλωτές σε ένα τυποποιημένο ενημερωτικό έντυπο για προσυμβατικές πληροφορίες. Αλλά δεν, είναι ικανο... δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη διαδικασία. Δεν υπάρχει ομοιόμορφο έντυπο, κάτι το οποίο αν υπήρχε θα ήταν πολύ θετικό και θα επιτρέπει τη μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. Αλλά δεν έχω δει κάτι στην πρόταση σε σχέση με την σύναψη σύμβασης, ακόμη και αν αυτή δεν συνοδεύεται από αυτό το τυποποιημένο ευρωπαϊκό έντυπο ε, ενημέρωση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή όταν ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί με βάση απαιτήσει οδηγία. θα πρέπει να ε, έχει κάποια προστασία ο καταναλωτής παρόλα αυτά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πώς παρουσιάζονται οι προσυμβατικές πληροφορίες. Θα πρέπει να είναι φιλικές προς τον καταναλωτή. Να είναι σαφής ε, ο πιστωτή θα πρέπει να εξηγεί όλους τους όρου της σύμβαση στον καταναλωτή, προτού συναφεί οποιαδήποτε σύμβαση πίστοσης. Γιατί όσοι δεν έχουν οικονομικές γνώσεις δεν θα πρέπει να είναι σε μειονεκτική θέση. Επίσης, προ διαφήμιση. Δεν έχουμε καταλάβει τι θα πει διαφήμιση για του στόχους οδηγία αυτή. Μπορεί το φαινόμενο να μην ήταν πολύ σοβαρό σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη όλοι είδαμε καταστροφικές επιπτώσεις λόγω ε, της σύναψης ανεύθυνων δανείων. Και αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια προληπτική προσέγγιση και να αποφύγουμε τέτοιες ε, πρακτικές που θα διδοθούν και θα θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών μα συστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μηχανισμό αξιολόγηση ε, ότι ο ε, δανειζόμενο μπορεί πραγματικά να πάρει αυτό το δάνειο και θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλέ ε, τα άτομα αυτά. Δεν θα πρέπει να πληγούν αρνητικά λόγω αφαιρεγκαιότητας ή λόγω αδυναμίας αποπληρωμής της πίστοσης. Ένα πολύ σημαντικό τελευταίο θέμα. Έχω αμφιβολίες σε σχέση με αυτό το σύστημα που βασίζεται στι απαιτήσει τη ε, χώρα καταγωγή. Νομίζω ότι δεν θα είναι ρεαλιστικό στην πράξη. Σω θα πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική λύση. Όπω παραδείγματο χάρη ελάχιστε απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλου ε, του ε, φορεί που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Uh, the Οι πράσινοι θέλουν να μιλήσουν. Εγώ είμαι σκιώδης, λέει κυρία Ρούλε, και με, πραγματικά με ενδιαφέρει και πολύ το θέμα αυτό. Ήδη συζήτησα και συνεργάστηκα με τον κύριο Λέχνερ στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη και το θέμα εδώ είναι παρόμοια και γι' αυτό ήθελα να είμαι σκιώδης. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό η οδηγία αυτή να περιοριστεί καταρχήν στα θέματα των καταναλωτών. Βέβαια εδώ συμφωνώ με τον προελίσαντα ότι συζητήσαμε επαρκώς ε, το θέμα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Ε, έχει δίκιο ο κ. Λέχνα σε ένα σημείο, ένα πολύ κεντρικό θέμα της ε, πίστης για την αγορά κατοικίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούν τα διάφορα εθνικά συστήματα. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά την αγορά ή την ενοικίαση κατοικία, το μέγεθος των κατοικιών, τα διαφορετικά συστήματα ε, πιστώσεων. Ορισμένες χώρες έχουν παράδοση πολύ μακροχρονίων πιστώσεων που έχουν μόνιμο, σταθερό επιτόκιο. Δεν πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά, θα υπήρχε σύγχυση. Και αν δούμε ποιε ήταν οι επιπτώσει τη χρηματοπιστική κρίση, βλέπουμε ότι ακριβώ εκείνε οι χώρε που έχουν μακροπρόθεσμη δέσμευση όσον αφορά το, την πίστοση αυτή, είναι εκείνε που είχαν τα λιγότερα προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν το σύστημά του και να μην τεθούν σε πίεση. Το πρόβλημα των πληροφοριών είναι ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, εκείνοι που χρειαζόνται τις περισσότερες πληροφορίες γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλη ιδέα του θέματος, δεν μπορούν να κατανοήσουν, ας πούμε, 20 σελίδες πληροφορίες. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές πληροφορίες και να τις υποβάλουμε κατά τέτοιο τρόπο στον καταναλωτή, ώστε είναι ευανάγνωστες και ευνόητες. Τέλο. Όσον αφορά την εξέταση της ε, φερεγιότητας, ε, συμφωνώ ε, ότι πρέπει να τα τα πράγματα, κύριε Λέχνερ. Χρειάζεται βέβαια κάποια διευκρίνηση, γιατί η ανεύθυνη χορήγηση πιστώσεων ε, οδήγησε σε προβλήματα όχι μόνο τη ΣΥΠΑ, ΕΕ, αλλά και την Ισπανία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνουμε με το θέμα της φερεγιότητας. Ευχαριστώ. you very much. next... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φόξ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον τη της νομοδότησης κύριο Λέχνερ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικό θέμα η συμβάση πίστοσης ε, ε, για την ε, ενία αγορά και επομένως θα πρέπει να θέσουμε πολύ ψηλά ε, πρότυπα. Ε, καταλαβαίνω την, ε, τον προβληματισμό του κυρίου Λέχνερ σχετικά με την συστηματική προσφυγή στις κατεξουσιοδότηση πράξης που μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα και βεβαίως το, το, το θέμα του κατά πόσον μπορεί κανείς να πάρει αυτή αυτό το δάνειο, αυτή την υποθήκη ε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Κατά την άποψή μου, εδώ η Επιτροπή έχει κάνει λάθος και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει λίγο την άποψή της. Έχω ε, τρία άλλα μελήματα σε σχέση με το ε, θέμα που μας απασχολεί και νομίζω ότι ο κύριος Λέχνερ μπορεί να τα συμπεριλάβει στην γνωμοδότησή του. Άρθρο 2 της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτά τα buy to let, ε, ε, αυτές οι buy to let ε, πιστώσεις, αυτές διαφέρουν πολύ από ένα καθαρά στεγαστικό δάνειο βάσει καθαρής στεγαστικής υποθήκης. Είναι μία επένδυση, είναι μία επιχειρηματική λύση και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται εδώ ίδιο ποσοστό προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, σχετικά με το άρθρο 17 λέμε ότι θα πρέπει η πληροφόρηση να αφορά ε, μία σειρά στοιχείων παρόντων στην αγορά. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι δανειστές ε, έχουν ε, δει ε, συμβάσεις οι οποίες είναι αντίστοιχες με αυτήν που προτίθενται να υπογράψουν, όχι οποιοδήποτε είδους σύμβαση. Επίσης, σε πολλές ε, χώρες μέλη δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί υποστήριξης ε, και, εν πάση περιπτώσει, ε, δεν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, κάνοντας ένα γενικό σχόλιο. Δηλαδή, ότι ενδεχομένως οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της ζωής τους πληρώνουν περισσότερο σε τόκους που αφορούν υποθήκες και στεγαστικά δάνεια περισσότερο από ό,τι πληρώνουν σε οτιδήποτε άλλο. Και επομένως θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι πιστώσεις αυτές να δίνονται με επιτόκια πιο φιλικά έτσι ώστε τελικά να μην οδηγούν στην οικονομική εξακρίωση των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεκινούμε έχοντας τις καλύτερες των προθέσεων. Τελικά όμως φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου ζημιώνονται πολύ οι καταναλωτές. Απ' την άλλη πλευρά, προσπαθώντας ενδεχομένως να προστατεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ίσως να επιβάλλουμε επιπλέον χρεώσεις και αυτού του είδους οι υποθήκες να γίνουν ακόμα πιο ακριβές. Πρέπει να προσέξουμε. Έχετε δίκιο, λέει η Πρόεδρος, έχετε δίκιο. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε. Η κυρία Ροϊτόβα. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Να ρωτήσω λοιπόν εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει κάποιες μελέτες ή αναλύσεις σχετικά με τις ουσιώδεις τροποποιήσεις ε, τις οποίες θα επιφέρει αυτή η οδηγία και κατά πόσον ε, θα υπάρξει καλύτερη προστασία των καταναλωτών και επίσης καλύτερη αντιμετώπιση των καταναλωτών από πλευρά των τραπεζών. Σε πολλές χώρες ε, δεν υπάρχει ε, το, η νομοθετική βάση έτσι ώστε να εφαρμοστούν ε, αυτού του είδους ε, τα μέτρα. Επίσης, ένα θέμα σχετικά με την εμβέλεια αυτής της οδηγίας. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις και θα πρέπει να τις δούμε. Συμφωνώ πάντως ότι οι καταναλωτές πρέπει οπωσδήποτε να επωφεληθούν εναρμονισμένης πληροφόρησης και να έχουν ας πούμε κάποια δυνατότητα τυποποιημένης πληροφόρησης. Και νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να αφήσουμε και κάποιο χώρο για εθνική ερμηνεία κατεξουσιοδότηση πράξη σε πολλά από τα άρθρα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί ενδεχομένως να είναι ε, να, να είναι κάτι λογικό. Άρθρο 11. Πιστεύω ότι εκεί υπάρχει μία έλλειψη σαφήνειας, καθώς επίσης και στο άρθρο 22 και επ' αυτόν θα ήθελα ε, ο εισηγητής κάπως να αποσαφηνίσει τα πράγματα. Κυρία Στήλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Όπως και άλλοι προείπαν, είναι μια μακροχρόνια δέσμευση η σύμβαση αυτής της πίστοσης και συνεπάγεται και τη μεγαλύτερη επένδυση και φυσικά και το μεγαλύτερο κόστος σε περισσότερες περιπτώσεις για τους καταναλωτές. Εάν δεν μπορεί να εξοφλήσει τις δόσεις, ε, ο ε, συμβαλόμενος έχει κάποιες φορές αυτό ως αποτέλεσμα ολόκληρες οικογένειες να μείνουν στο δρόμο, να χάσουν το σπίτι τους. Οι οικογένειες πολλές ε, υφίστανται πάρα πολύ σημαντικές οικονομικές πιέσεις, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το όλο θέμα αυτό. Μίλησαν διάφοροι για τον ανταγωνισμό, για την αγορά των συμβάσεων πίστοση. Σίγουρα οι καταναλωτές είναι σημαντικό να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιλογής ε, για να προβούν ε, στη σωστότερη επιλογή. Μια ανοιχτή υγιής αγορά είναι σίγουρα απαραίτητη. Άκουσα κάποιους να κατηγορούν ε, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιλογή και αυτό με εξέπληξε. Εγώ θα έλεγα ότι ε, κάποιες φορές ε, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγοραστές ε, πρώτης κατοικίας, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά πλέον. Άρα δεν φταίνει η, δεν φταίνει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φταίνει οι τράπεζες. θα πρέπει επίσης να δούμε και το θέμα της εμπορίας του μάρκετινγκ και της ενημέρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν κάποιο λαμβάνει ενημέρωση πριν από τη σύναψη τη σύμβαση, αυτή η ενημέρωση, αυτέ οι πληροφορίε θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερε και σαφέστερε, ώστε να μπορεί ο καταναλωτή ε, να συνειδητοποιήσει όλε τι συνέπειε είναι πολύ σημαντική η απόφαση που έχει να λάβει ο καταναλωτή. Επίση, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για κάποια σημαντικά ενημερωτικά έγγραφα. Νομίζω ότι η σαφή η πληρότητα και η ευληπτότητα των πληροφοριών είναι το σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την πρόορια αποπληρωμή, είναι πολύ σημαντικό. Ο εισηγητή είπε ε, και για το remortgaging, μίλησε για την αναχρηματοδότηση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και χαίρομαι που τα αναφέρατε. Τελευταίο ερώτημα προ την Κομισιόν. Πόσοι ε, πολίτες έχουν ε, αναζητήσει σύμβαση πίστοση σε μια άλλη χώρα από τη δική τους. Θα με ενδιαφέρει να ξέρω την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρός μας είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν ήθελα να επισέλθω ε, στην ουσία της συζήτησης γιατί ακούσατε τα σχετικά του σκιώδης Απλά θα ήθελα να μιλήσω για τη διαδικασία συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι στις συντονιστές ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε εμείς καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Αλλά ιστορικά ε, το υπόβαθρο ποιο είναι. Το θέμα είναι να έχουμε μια πιο ομοιογενή αγορά ε, στις υποθήκες. Και υπήρξε και πράσινη βίβλος στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ο Τζον Πέρβης που έχει πάρει σύνταξη ήταν ο αρμόδιος συνάδελφος από την Οικονομική Επιτροπή που είχε αναλάβει το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας όμως ε, είχε αποκλειστική αρμοδιότητα πράγματι για τις πτυχές προστασίας καταναλωτών αυτής της έκθεσης. Έχουμε προηγούμενο επομένως. Άρα ε, οι συντονιστές, για να σας απαντήσω και στο ερώτημα, θέλουν πραγματικά να ε, κρατήσουμε τις αρμοδιότητες που έχουμε και να έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένες πτυχές που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών. Όπως είπε και ο συγκητής, υπάρχουν κάποια παράλληλοι, υπάρχουν και τι παραλληλισμοί ε, για τις διατυπώσεις που αφορούν τις, την προστασία των καταναλωτών καταναλωτική πίστη είναι μια, ένας είχαμε την αρμοδιότητα σε επιτροπή, επομένως αυτό που θέλω πρώτα απ' όλα εγώ να κάνω είναι η δική μας Επιτροπή να εστιάσει στους τομείς για τους οποίους έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Ίσως να θέλουμε να σχολιάσουμε και άλλους τομείς ε, της πιθανής νομοθεσίας. Όπως προείπαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα κίνητρα ε, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, που στόχο είχε πολύ περισσότερο τη δημιουργία μιας ε, ενίας αγοράς, ενώ τώρα πιο πολύ σχετίζεται με την προστασία των καταναλωτών, γιατί είδαμε κάποιες πολύ κακές πρακτικές που οδήγησαν ε, πολλούς καταναλωτές ιδιαίτερη μειονεκτική θέση και βέβαια ε, προήλθαν από αυτά όλα αυτά τα φαινόμενα και όλα τα ζητήματα ε, με τις συνάψεις δανείων από τις τράπεζες και όλα τα επακόλουθα. Νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα έχουμε να επιτελέσουμε πολύ σημαντικό έργο σε αυτό το πλαίσιο ως Επιτροπή. Και τέλος, θα μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα, αλλά πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή να σας εξηγήσω. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομοσματικών Υποθέσεων έχει προσφέρει ενισχυμένη συνεργασία με μας. Αλλά όχι αρμοδιότητα αποκλειστική για οποιοδήποτε άρθρο. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ θα κάνω μια αντιπροσφορά όταν την έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα, η Οικονομική Νομισματική Επιτροπή προτείνει ένα πάρα πολύ μικρό, που δεν μπορούμε να δεχθούμε, πολύ σύντομο χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση έχει ε, συνταχθεί ήδη ένα χρόνο πριν, την, ε, πριν επιληφθούμε εμείς στο Κοινοβούλιο και υπάρχει και μια ακρόαση που προβλέπεται. Ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Η Επιτροπή μας να έχει τη δυνατότητα πραγματικά να εξετάσει τα στοιχεία που αφορούν την προστασία των καναλωτών. Θα σας πω την άποψη του Πρόεδρου. Ξέρω ότι οι συντονιστές και νομίζω όλοι είναι παρόντες, ε, στηρίζουν. Ε, ας δώσω το λόγο στην Πρόεδρο. Ας ακούσουμε την, την Επιτροπή τώρα. Thank you. Thank you very much for the... Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ για τα τόσο επικοδομητικά σας σχόλια. Η πρώτη αυτή οδηγία είναι το αποτέλεσμα αρκετά μακρών προπαρασκευτικών εργασιών που άρχισε με μια πράσινη βίβλο, όπως είπε ο κ. Σάρβο, το 2004 αν δεν κάνω λάθος και οδήγησε σε μια λευκή βίβλο που οδήγησε σε ακροάσεις, μελέτες, εργαστήρια, εργασίες ομάδων εμπειρογνωμόνων που τέλος κατέληξα στην πρόταση που έχουμε εδώ ενώπιον σήμερα. Ο στόχος της πρότασης είναι προφανώς να είναι ένα βήμα προς την άγουσα που θα ανοίξει τις αγορές για τις πιστώσεις ακινήτων. <clears throat> Ταυτόχρονα όμως προσφέροντας και εξασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών και μία υπεύθυνη συμπεριφορά δανεισμού και διαδεδότησης από όλους τους ενδιαφερόμενους. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην αγορά των συμβάσεων πιστώσεων για κινήτα. Καταρχήν η ε, έλλειψη ισορροπίας από τις δύο πλευρές. <clears throat> Η αγορά όμως ε, χαρακτηρίζεται και από προβλήματα διακανονιστικά ή μεσάζοντας παραδείγματος χάρη ή, ή ορισμένα άλλα Ινστιτούτα που ασχολούνται μόνο με την ε, ε, χορήγηση πιστώσεων για κίνητα δεν ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο από τον νομοθέτη. Και είχαμε παραδείγματο χάρη προβλήματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι σήμερα δεν έχουμε μία ενιαία αγορά. Και παρόλο που δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία για τον αριθμό των ε, δανείων που δίνεται με υποθήκες διαμεθοριακά, ξέρουμε ότι ο αριθμός είναι λίγο πολύ στα μηδέν. Χρειάζεται λοιπόν μία σειρά δημάτων για να φτάσουμε σε διαμεθοριακού τύπου πιστώσεις για Τα όμως έχουμε ένα προληπτικό μέσο κατά ανευθύνωση ευθύνων δανειοδοτήσεων από κάποιους. Και είδαμε στα κράτη-μέλη, όχι βέβαια στην κλίμακα που το είδαμε στη ΣΥΠΑ, αλλά κάτι παρόμοιο με εκείνου που δανείζουν σε διαφορετικό νόμισμα, χωρίς να ε, ε προδοποιούν για τον κίνδυνο της δοδενότησης σε ξένο νόμισμα ή παραδείγματο χάρη ε, δανειοδότηση χωρίς πραγματικό έλεγχο των εισοδημάτων του δανειστού και των ε, δυνατοτήτων που έχει να επιστρέψει το δάνειο αυτό. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για τις προτάσεις της ε, Κομισιόν. Προσπαθήσαμε να παραμείνουμε αναλογικοί και να παραμείνουμε σε ένα επίπεδο εναρμόνισης που την αποκαλούμε ή εναρμόνιση στοχός. ο, στόχο είναι αυτό που μα ενδιαφέρει. Ορισμένε χώρε θέλανε ένα μέγιστο εναρμόνιση για κάποια σημεία, όπω παραδείγματο χάρη η προσυμβασιακή ενημέρωση. Άλλες φορές όμως γνωρίζουμε το ποσοστό διακυσμά διακυμάσεων στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά τα καθεστώτα που ισχύουν και θα πρέπει να αφήσουμε τη δυνατότητα ευελιξίας στα κράτη-μέλη για να παραμείνουν στο σύστημα που έχουν, που είναι αρκετά αποτελεσματικό τις περισσότερες φορές. Ορισμένοι αναφέρθηκαν ότι θέλουν να είναι απόλυτα ευθυγραφισμένη η οδηγία αυτή με την οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Εμείς προσπαθήσαμε η πρόταση της Κομισιόν να βασίζεται καταναλωτών στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη, αλλά πολλές φορές σε κάποιες διακοιμάσεις ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. και εν μέρει η δική μας πρόταση πάει πιο μακριά από την οδηγία για την κατανοητική πίστη, παραδείγματο χάρη για τους μεσάζοντες, που είναι οι μόνοι μεσάζοντες ε, που δεν ελέγχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το κατάλληλο ελεγκτικό σύστημα. Αυτό αφορά μου όπως σας λέω μόνο τους μεσάντους για την κατανοητική πίστη. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η υποχρέωση της αξιολόγησης ευθυγραμμισμένου με το θέμα του υπεύθυνου δανεισμού σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή προτείνει σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης να αρνούνται το δάνειο. Εάν δεν γίνεται αυτό, τότε γιατί να γίνεται η αξιολόγηση της φερεγγιότητας του δανειστή. Ορισμένοι θεωρούν ότι αν ε, πούμε ότι σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος της έρευνας αφαιρεγιότητας Εάν υπάρχει και η υποχρέωση αυτό να ανηθούν το δάνειο, αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά ότι αν ο έλεγχο αφαιρεγιότητας είναι θετικό, υπάρχει υποχρέωση της χορήγηση του δανείου. Αυτό δεν είναι σωστό όμως. Επίσης, θεωρούμε ότι ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της πρόορης επιστροφής του δανείου. Παρόλα αυτά, τα συστήματα που υπάρχουν στα διάφορα κρατημέλη διαφέρουν πολύ τα μένα από τα δε. Και παρόλο που η οδηγία προβλέπει το δικαίωμα της επιστροφής πρόωρα του δανείου αυτού, αυτό ίσως πολλές φορές υπάρχει σε διάφορους όρους που αποφασίζουν να ορίσουν στην Εθνική Νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Πρόεδρος, με συγχωρείτε που σας ε, διακόπτω, αλλά έχουμε άλλο ένα θέμα. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το θέμα τώρα των επιπτώσεων της πρότασης. Εμείς προσπαθήσαμε να δούμε κράτος ανακράτο κράτο ποιες είναι οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, ορισμένες χώρες εκμεταλλευτήκαν τη μεταφορά των, της οδηγίας για την κατανολική πίστη και την διεύρυναν την οδηγία αυτή για να καλύψει και τις πιστώσεις ε, ε για κατοικίες, για κίνητα. Γι' αυτό είναι δύσκολο να γίνει ακριβή ανάλυση των επιπτώσεων σε κάθε Σα Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κύριε Λέχνερ, πραγματικά χρειάζεστε ε, λίγο χρόνο για να ολοκληρώσετε. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ε, ναι, ευχαριστώ. Θέλω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχήν ε, είμαι ευγνώμων για αυτά που άκουσα σχετικά με την αρμοδιότητα. Το είχα σημειώσει και ξέχασα να σας το πω στην εισαγωγή μου. Γι' αυτό. Ε, είμαι ευγνώμων προς τον πρόεδρο και ε, πραγματικά είναι σημαντικό αυτό για όλους. Σε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θα πρέπει να πούμε ότι εν ώψη και αυτών που ρώτησε η κυρία Ρόιτοβα ότι δεν πρέπει να έχουμε σφαιρική και γενική καθολική αλλαγή αλλά βήμα προς βήμα προς βήμα. Αυτή είναι η ζωστή άποψη πολύ σύνομα στο θέμα της φεργαιότητας. Εγώ δεν νομίζω ότι η χρηματοπιστωτική κρίση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την οδηγία αυτή ή να αποφευχθεί στο μέλλον. Γιατί αυτό ασφορά πολλά άλλα θέματα. Και ότι δεν τηρήθηκαν παραδείγματος κάνει και οι διατάξεις. Δεν θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία δεν υπήρχαν αυξημένες ε, ε, πτωχεύσεις ε, και επίσης το θέμα της φεργιότητας. Σωστό είναι αυτό. Ε, τώρα να πούμε, εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και γι' αυτό θα πάρει αυτό το δάνειο. Ακούει το λογικό, αλλά τι σημαίνει αυτό η τελευταία αναλύση. Εάν αυτός ο υπάλληλος φοβάται ότι μετά από 8 χρόνια, ας πούμε, ε, κάποιο δικαστήριο αποφασίσει ότι α, δεν έπρεπε να έχει καταλήξει σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Αλλά ε, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ε, ε ασφαλιστικές δικλείδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Κατά λίγο στο συμπέρασμα σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε και χρειάζονται κάποιε διευκρινήσεις που θα μπορούν να γίνουν μετροπολογικές. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λέχνερ. Βεβαίως ε, θα έχουμε και τις διαπραγματεύσεις με την ΕΚΟΝ. Προσπαθούμε καταρχάς να διαπραγματευτούμε το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι ε, σημαντικό. Λοιπόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε και στις 20 Ιουνίου να στείλουμε την ε, έκθεσή σας, την γνωμοδότησή σας μάλλον και για μετάφραση, να έχουμε τουλάχιστον μέχρι τότε την, ε, μια αρχή. Ακούσαμε ότι η ΕΚΟΝ θέλει να ψηφίσει στις 11 Ιουλίου για, την, ε, για το θέμα και όλο αυτό είναι απαράδεκτο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει βέβαια ότι θα καταλήξουμε σε κάποια ικανοποιητική ε, στάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κορχόλα γιατί ήταν αρκετά ευγενής έτσι ώστε να ε, προεδρεύσει Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε ακόμα ένα θέμα. Έχουμε τον κύριο Σαλβίνη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ε, μήπως θα μπορούσατε να είσαστε μάλλον σύντομος έτσι ώστε να γίνουν και κάποια αρχικά σχόλια και φυσικά θα έχουμε και την δυνατότητα αργότερα να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Θα ήθελα επίσης ε, ε, να πω ότι έλαβα επιστολή από τον κύριο Σέμιτα σχετικά με τον εναρμονισμένο τελωνιακό ε, κώδικα. Ε, θα καλύψω το θέμα αυτό όταν έρθει η ώρα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Σαλβίνη και την κυρία Κορχόλα, Ράκτη Σμιτ και ο υποφαινόμενος. Και η Χάιντι Ρούλε, όχι, όχι, όχι. Κάποιος άλλος από την ΚΟΕ ενδεχομένως, όχι. Έχουμε λοιπόν πέντε ομιλητές και 15 λεπτά, αλλά εδώ έχουμε και η κυρία Ράπτη. Ναι, ναι, ναι, είσαστε σκιώδης συγγήτρια έτσι κι αλλιώς. και ε, Σαμίσκη, Σαλβίνη, 15 λεπτά θα πρέπει να είσαστε όλοι πάρα πολύ ταχύς, Κύριε Σαλβίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, από τις 15 μου, από ε, τις 15 μου σελίδες που περάσω στις 2. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή, καθώς επίσης και τη γραμματεία της ε, ε αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς να έχουμε μια πρώτη συνάντηση με τους σκιώδες συγητές και μετά 16 Ιουνίου την ακρόαση, το hearing. τι να σας πω τώρα, σε δύο λεπτά τι να πω. Τέσσερα κύρια σημεία. Έχουμε λοιπόν την υλοποίηση του επικυροποιημένου ε, κώδικα, τελωνιακού κώδικα, ο οποίος ε, προφανώς ε, δεν θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο τέλος του 2011. Χρειάζεται λοιπόν μια αναβολή. Με ποιο τρόπο θα γίνει η αναβολή αυτή. Θα ήθελα να μου πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν συμφωνούν με την αναβολή αυτή και αν υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οι οποίες ιδιαίτερα ιδιαίτερως αντιτίθενται στην εν λόγω αναβολή. Να μας ε, δώσει λοιπόν την άποψή της η Επιτροπή. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε ε, να ε, έχουμε και ένα νέο όρο έτσι ώστε σταδιακά να αρχίσει η εφαρμογή κάποιων από τις διατάξεις του επικαιροποιημένου τελωνιακού κώδικα. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ είναι επίκαιρη η συζήτηση για τα τελωνία ε, ε, έτσι ώστε να υπάρξει ασφάλεια των προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν ε, στην εσωτερική μας αγορά και βεβαίως για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε μέσα από γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες να μπορούν να εκτελωνίζουν τα προϊόντα τους τα προστατεύοντας ταυτοχρόνως τους καταναλωτές από οποιαδήποτε προϊόντα παραχάραξης ή άλλα ακόμα σοβαρότερα ε, θέματα όπως ας πούμε τρομοκρατία κλπ. Πρέπει να δούμε να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε πραγματικά οτιδήποτε περνάει από τα τελωνία μας. Ε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε στα τελωνία οτιδήποτε μπορεί να είναι προϊόν παραχάραξης ή προϊόν επικίνδυνο, ουσία επικίνδυνη για τους ε, καταναλωτές. Πρόγραμμα δράσης για τα τελωνία είναι ένα από τα κύρια στοιχεία αυτού του επικαιροποιημένου ε, κώδικα Ξέρετε ότι συχνά ε, ε, βλέπουμε εναρμόνιση σε επίπεδο των 27 ε, και εδώ βλέπουμε ότι και η κοινή λογική και η αποτελεσματικότητα την οποία όλοι επιζητούμε μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα τελωνία θα πρέπει να αποτελέσουν ένα από τα εναρμονισμένα πεδία για, τους, για την Ευρώπη των 27 θέλουμε ε, οπωσδήποτε να υπάρχει αρκετός χρόνος έτσι ώστε να αξιολογήσουμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο. Ε, και να πω στα πρακτικά θέματα ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι αυτή η οποία θα είναι επίσης αρμόδια. Ε, βεβαίως η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αφού μιλάμε για τελωνία θα πρέπει, τελωνία, θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, τι κάνουν οι άλλες χώρες, τρίτες χώρες, χώρες εταίροι και μη Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σεβαστεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης ε, κυρίως όσον αφορά τις επερχόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες επί του θέματος αυτού. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα άλλο γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Βεβαίως είμαι στη διάθεση όλων και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Well, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλβίνη. Πλούσιο στο περιεχόμενο και συνοπτικό στην παρουσίαση. Άρα προσβλέπω με και στην έκθεση που θα συντάξετε στο μέλλον. Σύντομε σκέψει από του Κιώδη θα ακούσουμε για τα συστήματα που θα θέλετε να λάβει υπόψη συγητή και έχει και συνεδρία των ε, σκιωδών σύντομη. Κυρία Κορχόλα είναι η πρώτη ομιλητρία. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχουν υπάρξει κάποιες δικαστικές βελτιώσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί και η συνεργασία των καλωνιακών ε, υπαλλήλων και των αρχών επιτήρησης της αγοράς. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και νωρίτερα όταν είχαμε μιλήσει για την επιτήρηση της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων. Αν εργάζεται αποτελεσματικά η πτήση αγοράς, αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει και στην δημιουργία ενός ισότιμου ε, πεδίου ανταγωνισμού γιατί κάποιοι φορείς μπορεί να έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα εάν τηρούν τις ε, διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι σε άλλες χώρες. Θα μπορούσαν, παραδείγματο χάρη, όταν έρχονται τα προϊόντα ε, στους λιμένες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε ε, έλεγχο και να έχουμε και μια ενισχυμένη συστηματική συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών υπαλλήλων και των υπεύθυνων επιτήρησης αγοράς. Αυτό είναι το βασικό που θέλω να πω. Ευχαριστώ. Mrs. Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη με τρεις λέξεις. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή, ο οποίος μας έδειξε το σωστό δρόμο πώς μπορούμε να είμαστε σύντομοι και ταυτοχρόνως περιεκτικοί. Ε, σκέπτομαι ότι το πρώτο ζήτημα είναι ο χρόνος. Χρειαζόμαστε χρόνο και ήταν, είναι κάτι το οποίο το ξέραμε από την αρχή. Όταν έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για τον εξυγχρονισμό του κανονισμού για τη λειτουργία των τελωνίων, είχαν τότε επισημανθεί ζητήματα που είχαν σχέση με το χρόνο. Ότι κάποιες χώρες, αρκετές χώρες θα είχαν πρόβλημα να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε σχέση με τα ηλεκτρονικά συστήματα. Άρα μια πρώτη μου σκέψη είναι ότι συμφωνώ με το χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφαλώς συνεργασία. Ε, άλλα δύο ζητήματα θέλω να βάλω, μερικές σκέψεις. Το ένα είναι η χρηματοδότηση και μιλάω για τη χρηματοδότηση και από την πλευρά των κρατών μελών και από την πλευρά της Κομισιόν ο, κυρίως στο θέμα του να έχουμε ένα περισσότερο αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα. Τελευταίο άφησα το θέμα του ελέγχου. Α, σκέπτομαι ότι ασφαλώς θέλουμε έλεγχο, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Αλλά από την άλλη μεριά σκέπτομαι ότι ε, πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή το θέμα του ελέγχου, ώστε να μην δημιουργήσουμε ε, ανάποδα αποτελέσματα. Ε, τι εννοώ, κλείνοντας με δύο κουβέντες. Ε, φτάσουμε σε υπερβολές που θα έχουν ως αποτέλεσμα πάρα πολύ πρακτικά να συσσωρεύονται τεράστιοι όγκοι εμπορευμάτων και κατά συνέπεια να μην λειτουργεί με την ταχύτητα που πρέπει η αγορά. Ε, αυτά μέχρι τώρα και προσβλέπω στην συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους χειώδεις για να βγάλουμε κάτι καλό ε, έχοντας πάντα στο μυαλό μας το όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Uh, κύριε Σμιτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λάθος κάνω που θα πω ότι το θέμα αυτό είναι υψηλής πολιτικής σημασίας και τις τελευταίες εβδομάδες ε, ακόμη περισσότερο. Δεν νομίζω να ασφάλω, διότι η τελωνιακή έλεγχη πλέον χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο. Επομένως, φυσικά και θα πρέπει να σκεφτούμε και για το χρονοδιάγραμμα. Είναι σόφρον και λογικό να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο ή μήπως αντιθέτως θα έπρεπε να αντιδράσουμε και να πούμε δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Γιατί αν δεν το αντιμετωπίσουμε, αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, ίσως θα έχουμε προβλήματα σε άλλους τομείς η αποτελεσματικότητα φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπημένη προσέγγιση, γιατί χρειάζεται να δράσουμε τάχιστα, κατά την άποψή μου. Δεν έχω τίποτε κατά σε σχέση με τα όσα είπε ο εισηγητής. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τώρα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, το ζήτημα είναι πάρα πολύ ε, πιο ζέων, θα έλεγα, από πολιτικής πλευράς σε σχέση με ορισμένε εβδομάδες πριν. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε, δεν θέλει το λόγο. Να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σαλβίνο, νομίζω ότι εντόπισε ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία. Θα ήθελα να ενισχύσω κι εγώ να πω για την υλοποίηση των ορισμένων του Κώδικα και όλα τα συστήματα πίσω από αυτόν. Όσοι είμαστε στην παρουσίαση εκ μέρου ε, τη ομάδα του κυρίου Σεβέτα, ίσω τα πει ο κύριο Αλέσκη, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα για την ετοιμότητα των κρατών μελών να υλοποιήσουν τον οργανισμένο κώδικα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα υπάρξει βέλτιστη δυνατή υλοποίηση και άλλο βέβαια θέμα και το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, κατά πόσον είναι ή όχι ρεαλιστικό. Κύριο Σεμέτα με επιστολή του επιβεβαιώνει ότι ακριβώς αυτό θέλει να κάνει η οχι ρεαλιστικο κυριο σεμετα με επιστολη του επιβεβαιωνει οτι ακριβώ αυτο θελει να κανει η κομισιον Θα το διανύμω ε, το γράμμα αυτό στα μέλη τη Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε και στην πρόταση του κυρίου Σεμέτα. Θα το κάνουμε επισήμω, θα το συζητήσουμε όμω. και ελπίζω η Κομισιόν να συμφωνήσει γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει μια στρατηγική συζήτηση για την υλοποίηση των νέων αυτών εργαλείων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ήδη βλέπουμε να υπάρχει μια σημαντική επανεξισορρόπηση των δραστηριοτήτων του τρόπου εργασία του Συμβουλίου και γενικότερα εντός Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσονται κάποια συστήματα για την ε, εισπράξη εσόδων και για την επεξεργασία εισαγωγών-εξαγωγών από πλευρά τη δημόσια πολιτική, όπω είπατε, πράγματι, νομίζω όλοι σα το είπατε άλλωστε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των προϊόντων. Έχουμε όμω και τα ζητήματα απομίμηση, απομιμήσεων, παραποιήσεων, που ε, είναι και στον πολιτικό κατάλογο προτεραιοτήτων. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο. Τι ρόλο θα έχει σε αυτή την όλη διαδικασία. Και τέλο, συνεργασία. Όταν ε, Πήγα πρόσφατα ε, και παρακολούθησα μια πολύ σημαντική επιχείρηση η οποία στέλνει εμπορεύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα ότι όλες οι αποστολές ε, ουσιαστικά γίνονται τη νύχτα και ο εκτελονισμός, τέλος πάντων, τελωνικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί στη διάρκεια της ημέρας. Και αυτοί που τα εμπορεύματα που σταματώνται είναι αυτά τα οποία ήδη είχαν εντοπιστεί πριν από την ανάλυση και από την εξολόγηση επιπτώσεων. Τώρα λοιπόν Μιλάμε για ε, πληροφορίες που συλλέγονται εκ των προτέρων και για αναλύσεις οι οποίες γίνονται εκ των προτέρων και όχι τη στιγμή της αποστολής. Δεν γίνεται μια κλειστή έτσι, εγκρυπτό και παραβίαση τα ανταλλαγή πληροφοριών, γίνεται εκ των προτέρων συλλογή των πληροφοριών και ανάλυσή τους. θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε αυτή τη ε, διαδικασία ανταλλαγής ε, πληροφοριών για να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι ομιλητέ, γι' αυτό θα παρακαλέσω τον κύριο Σαλέσκη να μας πει δύο-τρία πράγματα κι αυτός. Γιατί συναντηθήκαμε πριν από κάποιες εβδομάδες και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαλβίν και θα συζητήσουμε και το χρόνο διά... Όχι, σας, ε, μάλλον δεν είπα σωστά το όνομά σας, τέλος πάντων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί διαβλέπουμε εδώ ε, την δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου των τελωνίων και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στα πιο ε, σημαντικά. Τελωνιακός κώδικας. Ναι, πρέπει να πω ότι εμείς δεν θέλουμε να περιμένουμε την, ε, δεν περιμένουμε μάλλον την, τον εξυγχρονισμό ε, του τελωνιακού κώδικα. Κάθε μέρα εφαρμόζουμε ε, τα πάντα. Κάθε μέρα έχουμε νέα πρότυπα για ασφάλεια και επίσης έχουμε ενσωματώσει και το νέο κανονισμό IPR. Βεβαίως το NCC είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στενή συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των χωρών μελών έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ε, σύστημα πληροφορικής το οποίο θα είναι σε θέση διευρωπαϊκά ε, να ε, στηρίξει την, τα τελωνία. Μεγάλη συνεργασία βεβαίως μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι προϋπόθεση εκ των Προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τα κράτη-μέλη έτσι ώστε ώστε ε, να υπάρχει ένα ενιαίο πεδίο δράσης για όλους τους εμπορευόμενους. Καλωσορίζουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά την πρόταση και δηλώνουμε ότι είμαστε απολύτως στη διάθεση του εισηγητού κυρίου Σαλβίνη έτσι ώστε και βεβαίως και των υπόλοιπων μελών ε, για πλήρη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλενσκή. Κύριε Σαλβίνη. Θέλετε να πάρετε το λόγο, να πείτε κάτι για να κλείσουμε τη συζήτηση, να πείτε κάτι για την ακρόαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την επόμενη εβδομάδα με τους συγκιώδεις συγητές βεβαίως ε, θα ε, καθορίσουμε το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα ε, και να καθορίσουμε και τις έντες λεπτομέρειες ακρόασης που προβλέπεται αν δεν κάνω λάθος το πρωί της 16ης Ιουνίου. Βεβαίως θα, δώσω, θα στείλω σε όλους το γραπτό κείμενο της αρχικής μου παρέμβασης που λόγω στενότητος χρόνου δεν κατάφερα να διαβάσω έτσι ώστε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης και για την μελλοντική μας συζήτηση και βεβαίως θα πρέπει να λύσουμε και κάποια πολιτικά ζητήματα ε, έχουμε δουλειά μπροστά μας γι' αυτό να ξεκινήσουμε να ανασκουμποθούμε λέει ο μιλητής γρήγορα να ξεκινήσουμε άμεσα και να προετοιμάσουμε φυσικά και την ακρόαση της 16ης Ιουνίου. Μέχρι το απόγευμα θα έχουν όλοι και οι συνάδελφοι το κείμενο, το γραπτό κείμενο το οποίο είχα προετοιμάσει. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much Ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά παίρνετε πολύ σωστή θέση. Ναι, 5η 16 Ιουνίου, 10 με 12.30 το πρωί. Ε, ε, θα έχουν την δυνατότητα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βλέπουν στο διαδίκτυο και να ακούν στο διαδίκτυο το, ε, την ακρόαση αυτή. Και επίσης να σιγουρευτούμε ότι όλοι οι, όλες οι αρμόδιες αρχές ε, θα γνωρίζουν ότι κάνουμε την ακρόαση αυτή έτσι ώστε να μπορούν και εκ των υστέρων να στείλουν ε, και τα ε, σχόλιά τους. Λοιπόν, το αρχικό μας πρόγραμμα είναι προθεσμία κατάσταση των 20 Σεπτεμβρίου και θα το ξανασυζητήσουμε βέβαια το θέμα ολοκληρώσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα και θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων πάρα πολύ σημαντική ε, όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το απόγευμα και βεβαίως θα έχουμε και μία μήνυα ακρόαση η οποία θα ξεκινήσει στις 4 και θα αφορά τον εξυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι.